Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί σύμβουλοι, συνεργάτε, εκπρόσωποι τη βιομηχανία και πανελιστ. Σα καλωσορίζω όλου, με πολύ μεγάλη χαρά σα βλέπω στην Επιτροπή μας ε, στην ακρόαση ε, για τη βιομηχανία 4.0. Προηγουμένω όμως θα πρέπει και θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη αν δεν έχετε άλλα σχόλια μπορεί να θεωρηθεί εγκεκριμένη χωρίς αλλαγές σήμερα σε διάταξη. Δεν ξέρω, έχετε εσείς σχόλια. Δεν βλέπω να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Με μεγάλη θλίψη σας ενημερώνω ότι ο συνάδελφος Τζαλούκα Μπουονάνο έχασε τη ζωή του στις 5 Ιουνίου στην Ιταλία. Είναι πραγματικά πάρα πολύ θλιβερή αυτή η ιστορία. Ορισμένοι από εσά θα τη γνωρίζετε Φαντάζομαι θα μάθατε τα δυσάρεστα νέα. Ο κύριος Μπονάνο υπηρέτησε ως μέλος της Επιτροπής μας ΙΤΡΕ ε, από το 2014 που εξελέγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή για μια διετία. Ήταν μέλος ε, της ομάδας ε, «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας». Πριν εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διετέλεσε μέλος της Ιταλικής Βουλής από το 2008 έως το 2000. 14. Επί μία εξαετία ω πρόσωπο του κόμματο Λέγκα του Βορρά Λέγκα Νόρτ. Αφήνει πίσω του γυναίκα και δύο παιδιά, Στου οποίου θα ήθελα να ε, απευθύνω τα πιο ειλικρινή συλληπιτήρια εξ ονόματο όλων των μελών τη επιτροπή μα. Θα σας πρότεινα στην αρχή της συνεδρίασης λοιπόν να τηρήσουμε ένας λεπτού σιγή στη μνημή του συναδέλφου μας κλεπώντος μέλλοντος της Επιτροπής, ε, μέλους, συγγνώμη, της Επιτροπής Thank you very much. Σε ευχαριστώ πολύ. Uh, λοιπόν, θα ήθελα να σας θυμίσω επίσης ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ως προς τις προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών για τα εξής θέματα θα είναι πολύ σημαντικό για πολλούς από εσάς. Πρώτον, το ραδιοφάσμα, οι συχνότητες, η συγκεκριμένη είναι η κυρία Τόγια, νέα προθεσμία, είναι η 1η Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Μαντί, για την 30η Ιουνίου παρατάθηκε κατά 24 ώρες. Καμιά φορά αυτό είναι απολύτως αποφασιστικό, διότι συνήθως τελευταία στιγμή καταθέτουμε τις τροπολογίες. Έχουμε πάρα πολλέ τελευταίε στιγμέ ακόμα. Ανταλλαγή πληροφοριών, μηχανισμό, δηλαδή στην ενέργεια για την ανταλλαγή πληροφοριών ε, μεταξύ των κρατών μελών Καστοντεύσκη, 1η Ιουλίου, 12 το μεσημέρι, το, αυτό αντί για τις 30, δηλαδή, Ιουνίου. Θα αλεί και mail με όλες τις αλλαγέ, προς όλα τα μέλη. Λοιπόν, τώρα περνάμε στην ακρόασή μα. Είναι το σημείο 3 για δημόσια αγρόση με θέμα εξετάζοντα τη βιομηχανία 4.0 σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο τη ρομποτική και των μαζικών δεδομένων επί τη βιομηχανία. Τα λεγόμενα big data είναι αυτά. Καλωσορίζω τους ομιλητές μας. Με πολύ μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε όλους ε, σήμερα ενώπιον μας. Το θέμα είναι άκρος σημαντικό βεβαίως ε, για την Επιτροπή μας και από τη δική μας σκοπιά, διότι είμαι θα, ε, αρμόδιοι και ε, για τη βιομηχανία. Όχι μόνο τι μεγάλε και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, αλλά και για την ψηφιακή ένωση, το ψηφιακό θεματολόγιο, τη ψηφιακή εσωτερική αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις πλατφόρμες, βιομηχανίας και όλα αυτά που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, περί τη ψηφιακή ένωση. Είναι το ο πιο Σημαντικό φάκελο, α πούμε η ψηφιακή ένωση, όχι μόνο η ψηφιακή εσωτερική αγορά. Θα ήθελα επίση να προσθέσω ότι η βιομηχανία 4.0 έχει πολύ μεγάλη επιρροή στη ε, διαδικασία βιομηχανική παραγωγή. Έχουμε διάφορε μορφέ τεχνολογίας, τα ε, μεγάλα μαζικά δεδομένα, τη ρομποτική, αλλάζει τελείω ε, η παραγωγή. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε και τα διάφορα σενάρια, το δυναμικό που ανοίγεται και ενδεχομένω την απαιτούμενη νομοθεσία. Αυτό είναι για μας το ζητούμενο και το σημαντικότερο ε, και θέλουμε να ρωτήσουμε όλους τους ομιλητές αυτής εξ αρχής. Χρειάζεται ε, νέα νομοθεσία. Τι χρειάζεται, σε ποια κατεύθυνση και θα θέλαμε να μας δώσετε τα φώτα σας και κάποια καθοδήγηση από πλευρά σας, έτσι όπως το βλέπετε εσείς, ειδικοί για τα θέματα μαζικών δεδομένων επίσης μας ενδιαφέρουν τα μάλλα. Είναι πολλές οι εκθέσεις στην Επιτροπή μας, ε, την Επιτροπή Ήτρε, που ασχολούνται ε, και είναι ε, πολύ συναφείς με το ρόλο αυτή της βιομηχανία, τα θέματα της ψηφιακής, ας πούμε αστικό δίκαιο και ρομποτική ή προς μία πράξη για την ενιαία ψηφιακή αγορά, η πρωτοβουλία για το ευρωπαϊκό cloud πριν από λίγες μέρες. Θα ακούσουμε όλους τους ομιλητές μας λοιπόν και στη συνέχεια μετά τις τέσσερις ομιλίες θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα παρακαλούσα τους ομιλητές μας να τηρήσουν το χρόνο που τους έχει δοθεί δεκάλεπτο. Θα έχετε την ευκαιρία και μετά το τέλος της συζήτησης, αν θέλετε, να προσθέσετε οτιδήποτε άλλο απαντώντας στις ερωτήσεις, συνοψίζοντας, θα έχετε τη δυνατότητα να δευτερολογήσετε, που μπορεί να είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα η δεύτερη τοποθέτησή σας για τα μέλη. Θα παρακαλούσα λοιπόν να τηρήσετε το χρόνο σας. Και αν μου επιτρέπετε, να δώσουμε το λόγο στον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Ματίας Πουτς, που είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Φρανχόφερ για εργαλειομηχανές και ε, για την τεχνολογία κατασκευών. Είναι μηχανολόγος. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Ε, αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και εργάστηκε και στο Λονδίνο το ε, μέχρι το 1994 ε, σε ένα δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου. Ο καθηγητής έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και βιβλία για το cloud computing, για την ε, ε, βιομηχανία 4.1. Αλλά διαβάζω λάθος βιογραφικό, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, στο Πολυτεχνείο του Χέμνιτς έχει σπουδάσει ο κύριος που Συγγνώμη, έκανα λάθος στον ομιλητή. Και βεβαίως ε, έχει και διδακτορικό και ε, είναι στο Ινστιτούτο Φρανχόφερ από το 1994. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά, κύριε Ματίας Πούτς, έχετε το λόγο ως πρώτος ομιλητής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για τις δικές μας ε, ιδέες. Εγώ είμαι μηχανολόγος, μηχανικός και στη Γερμανία έχουμε μία πραγματική παραγωγή μέσα στα πλαίσια της εργασίας του Ινστιτούτου μας. Ασχολούμαστε με τις ε, εργαλειομηχανές, forming technology και κάθε χρόνο κάνουμε έρευνες στον τομέα της βιομηχανίας. Αν μιλήσετε για τη βιομηχανία 4.0, το θέμα είναι ευρύτατο και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μεταφορά δεδομένων και τα ε, πρότυπα, τα business ε, models. Εγώ θα σας μιλήσω για το εργοστάσιο. Θα ήθελα να με παρακολουθήσετε με τη φορά του ρολογιού ε, με την εικόνα που βρίσκεται πάνω-πάνω για να δείτε από πού προέρχονται τα υλικά και τα υλικά αυτά εμπεριέχουν όλα τα δεδομένα και στη συνέχεια μπαίνουμε σε επεξεργαστές που ξέρουν τις παραμέτρους, τη λειτουργία και μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο, μια μεμονωμένη διαδικασία, πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και μπορούμε να προσαρμοστούμε με βάση τα δεδομένα. Έχουμε ψηφιοποίηση με βάση την χρήση που, τη χρήση των εργοστασίων έτσι ώστε να υπάρξει βελτιστοποίηση. Και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μία διάδραση μεταξύ όλων αυτών των προτύπων. Χρησιμοποιούμε την ενέργεια, το, τους διάφορους συγχρονισμένους πόρους και τα υλικά από τους διάφορους τομείς και έτσι φτάνουμε στο τελικό προϊόν γνωρίζοντας την ιστορία ε, του κάθε δεδομένου. Εδώ πρόκειται για μια πραγματικότητα, δεν πρόκειται για μελλοντολογία. Το κάνουμε εμείς, μπορούμε να το κάνουμε οι Κινέζοι, μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Το κάνουμε μέσα στα πλαίσια μίας πορείας με τη ε, φορά του ρολογιού. Αλλά δεν υπάρχει διασύνδεση πάντα των δεδομένων. Πρόκειται για στοιχεία, για δεδομένα και από τα δεδομένα φτάνουμε σε πληροφορίες, μετά φτάνουμε σε γνώση και στη συνέχεια σε προστιθέμενη αξία. Είναι λίγο περίπλοκο, αλλά εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω περισσότερο για το τι γίνεται σήμερα η βιομηχανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα τελικά δεδομένα. Δεν παράγουμε εμείς τα δεδομένα, τα αναλύουμε και δημιουργούμε την πληροφορία. Εμείς είμαστε χρήστες και εγώ πιστεύω ότι εάν τα δεδομένα είναι ε, πηγή καινοτομίας για το μέλλον, θα πρέπει τα δικά μας προϊόντα, οι δικές μας μηχανές, η τεχνολογία, τα υλικά μας να βρίσκονται στην εμπροστοφυλακή της ροής δεδομένων. Έχουμε παραδείγματα γι' αυτό. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά projects στο Ινστιτούτο μου ασχολήθηκα με ε, ένα θέμα όπου συλλέγουμε δεδομένα από τις εργαλειομηχανές, τα χρησιμοποιούμε, τα καταγράφουμε και παράγουμε στοιχεία έτσι ώστε να έχουμε αποθήκευση δεδομένων, μια ε, διαδικασία διαγνωστικής και συντήρηση. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε και μηχανές ε, βοήθειας στη χρήση ως προς την κινητή τηλεφωνία, τις ταμπλέτες και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να έχουμε τη σωστή πληροφορία την σωστή χρονική στιγμή. Και αν βρισκόμαστε κάπου μεταξύ, δηλαδή της φυσικής πραγματικότητας και του κυβερνοχώρου, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τους εργαζομένους στο εργοστάσιο και πιστεύουμε ότι θα έχουμε να κάνουμε με ένα μέλλον της κοινωνικής βιομηχανίας όπου θα έχουμε δίκτυα προστιθέμενης αξίας. Θα είναι κοινωνικά δεδομένα και μεταδεδομένα. Μιλάμε για τρεις έννοιες όπως βλέπετε στη διαφάνεια και στην τρίτη περίπτωση θα ήθελα να σας πω ότι βρισκόμαστε ήδη στη ρομποτική και γι' αυτό μιλάμε για την αξιολόγηση, για την εργονομία, αλλά και για θέματα αισθητήρων και ούτω καθεξής και θέματα αποδοχής. Εδώ ως παραγωγή πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η διάδραση ανθρώπου με ρομπότ στα ε, θέματα επικοινωνίας και αποδοχής. Τέλος, θα ήθελα να σας δώσω δύο εικόνες. Η παραγωγή Good Feeling. Αριστερά, όταν είχαμε τη βιομηχανία 0, 0 τότε στην εποχή της ε, Πέτρας προσπαθούσαμε να βρούμε μία αλληλεπίδραση δεδομένων χρησιμοποιώντας ή τρίβοντας τις δύο πέτρες. Επίσης, στη συνέχεια, στα πλαίσια της βιομηχανίας και των εφαρμογών προσπαθήσαμε να δούμε αυτό τον αλληλοσυσχετισμό. Φτάσαμε λοιπόν στο 1.0.2.0 και 3-0 και δεν θέλουμε να υπάρχει αυτός ο πολυσχηδής χαρακτήρας πάντα. Θέλουμε να υπάρχει εξειδίκευση και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να ευεργετηθούμε από την πολυπλοκότητα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο ευεργέτημα της βιομηχανίας 4.0. Το σύστημα είναι περίπλοκο, έχουμε πληροφορίες και θα έχουμε τις πληροφορίες και οι φυσικοί νόμοι δεν μας αποτρέπουν από κάτι τέτοιο. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πολυπλοκότητα για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τα μεγάλα και τα μικρά δεδομένα που μας παρέχει η ευρωπαϊκή κοινότητα. Μιλάμε όμως για τις κατασκευές. Δείτε για παράδειγμα αυτό το πολύ απλό στοιχείο. Σε σχέση με τη χρήση των ε, ρουλεμάν ξέρουμε πώς ε, έχει η παραγωγή και όταν βλέπουμε το κύκλο ζωής, τη χρήση, βλέπουμε ποια είναι τα δεδομένα. Αν δείτε λοιπόν αυτό το ρουλεμάν με τα διάφορα εξαρτήματά του, δεν θα ήταν σκόπιμο να δούμε πώς μπορούμε να παράγουμε στοιχεία όχι με επιπρόσθετους αισθητήρε, αλλά χρησιμοποιώντας τις ε, ε, γνώσεις μας με βάση την ανοτεχνολογία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, παράγουμε στοιχεία. Και δεν δε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά στα δικά μας δεδομένα ξεκινώντας με τα δεδομένα, στην πληροφορία, μετά στη γνώση και στη συνέχεια στο τελικό προϊόν. Δηλαδή θα πρέπει να παράγουμε στοιχεία και να μην φοβόμαστε την ε, περιπλοκότητα. Γιατί αυτά τα στοιχεία δεν θα μπορούσαν να παραχθούν σε άλλα σημεία του κόσμου που μας ανταγωνίζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρώτη τοποθέτηση και παρουσίαση της ακρόασή μα. Θέτει και φιλοσοφικά ζητήματα και ερωτήματα. Θέμα της αποδοχής, ε, πώς αισθάνεται κανείς όταν παράγει, πώς συνεργάζονται τα ρομπότ με τους ανθρώπους, πάρα πολύ σημαντικό και για τη δική μας Επιτροπή, τα κοινωνικά δίκτυα και ο κλάδος ε, πώς μπορούμε να υποφεληθούμε από την περιπλοκότητα, την πολυπλοκότητα. Δεν είναι πάντα κάτι το αρνητικό που θα πρέπει να φοβόμαστε και πώς ε, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα ερωτήματα που εθέσατε. Προφανώς δεν έχετε όλες τις απαντήσεις, αλλά πολλές ερωτήσεις έχουν και οι συνάδελφοι, οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά. Δεύτερος ομιλητής είναι ο κύριος Πέτερ Μπρόιτιγκαμ ε, που είναι από το δικηγορικό γραφείο ΝΟΕΡ. Εκείνος είναι απομοφητής από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, δικηγόρος και έχει εργαστεί στο Λονδίνο σε δικηγορική εταιρεία, όπως σας είπα προηγουμένως. Έχει γράψει δε σειρά ε, δημοσίευσεων και έργων για την βιομηχανία 4.0, για το cloud computing, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα πάντα είναι της αρμοδιότητας της δικής μας Επιτροπής. Είστε ακριβώς στον κατάλληλο τόπο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι προνόμιο για μένα να μπορώ να μιλήσω σε εσάς. Πού είναι διαφανής μου όμως. Μάλιστα, ωραία. Είναι βαρετό το θέμα, δίκαιο, αλλά τι να κάνουμε είναι σημαντικό. Γιατί γνωρίζετε ότι οι δικηγόροι πάντοτε έρχονται σε επαφή με τους ε, τεχνίτες και τους επιστήμονες ε, και μπορεί να υπάρχουν κάποια άλλη τα ζητήματα που χρήζουν ερμηνεία. Ε, και ιδίω για τη ρομποτική και τα μαζικά δεδομένα έτσι είναι η κατάσταση. Ας δούμε πρώτα τη ρομποτική και να δούμε τα ζητήματα της ευθύνης, το liability. Χρειάζεται εδώ ρύθμιση. Το επόμενο σημείο είναι το e-person. Δηλαδή χρειαζόμαστε κάτι τεχνητό, ειδικό, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα ρομπότ, ένα ηλεκτρονικό πρόσωπο, λοιπόν, για να έχουμε μια ευθύνη για το ε, ρομπότ που δεν θα είναι ε, μόνο πλέον τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και τα ρομπότ. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο ορισμό. Και το τρίτο Θέλω να συμφωνήσω απολύτω με τον προλαλήσαντα. Τα big data, τα μαζικά δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει εδώ να ρυθμίσουμε κάτι ή αρκεί η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Ας δούμε λοιπόν ένα-ένα τα θέματα αυτά. ability ευθύνη. Θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των πραγματικά αυτόνομων προϊόντων αφενός και των αυτοματοποιημένων προϊόντων αφετέρου. Δείτε τα αυτοκίνητα. Στα αυτοκίνητα υπάρχουν συστήματα υποβοήθηση τη οδήγηση, βοηθούν τον οδηγό να σταθμεύσει, να βρει το δρόμο του, να κρατάει τι αποστάσεις, αλλά παρόλα αυτά ο οδηγό εξακολουθεί να είναι αυτός που πρέπει να οδηγήσει. Δεν υπάρχει αλλαγή. Αυτά είναι τα αυτοματοποιημένα συστήματα. Στο μέλλον όμω και όλοι το συζητούν, θα έχουμε πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα οχήματα, ένα αυτόνομο ρομπότ που θα τα κάνει όλα μόνο του, θα πάρει αυτό όλες τις αποφάσεις, άρα ο οδηγός δεν θα παρεμβαίνει καθόλου και μάλιστα δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει γιατί το ρομπότ θα τα κάνει καλύτερα από τον οδηγό. Αυτό θα πει αυτόνομη οδήγηση, αυτόνομο σύστημα. Και αν δούμε τώρα την ευθύνη για τις αυτοματοποιημένες αυτές υπηρεσίες, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται νέα νομοθεσία η ισχύουσα νομοθεσία αρκεί. Αν δείτε την ευθύνη για τα προϊόντα, ιδίω την ευθύνη του, του κατασκευαστή, αρκεί. Γιατί τελικά τον έλεγχο τον έχει ο άνθρωπος, ο ίδιος ο κατασκευαστής. Δεν είναι self-learning. Για τα αυτοκίνητα επίσης νομίζω το σύστημα που ισχύει αρκεί. Έχουμε την ευθύνη του οδηγού του καταχωρημένου ιδιοκτήτη και του κατασκευαστή. Τρία πρόσωπα. Και αρκεί αυτό πιστεύω. Αν τώρα τα δικαστήρια ε, ερμηνεύουν όλο και πιο αυστηρά τον νόμο, είναι μια τάση αυτή που υπάρχει πράγματι στα συστήματα. Για τα αυτοματοποιημένα προϊόντα, τελικά ποιος αποφασίζει ε, στην τελική ανάλυση ο άνθρωπος και η φυστάμενη νομοθεσία νομίζω ότι είναι επαρκής, αλλά για τα πραγματικά αυτόνομα συστήματα, self-learning systems, εκεί το σύστημα δεν το ελέγχει ο άνθρωπος πλέον, ε, τα συστήματα λαμβάνουν μόνο τους τις αποφάσεις. Επομένως εκεί υπάρχει ένα κενό κατά την άποψή μου. Όταν λοιπόν φτάσουμε πραγματικά σε αυτά τα αυτόνομα συστήματα θα πρέπει να επανεξετάσουμε την νομοθεσία και ίσως τότε να εστιάσουμε σε τρία πρόσωπα. Στο χρήστη, στον κατασκευαστή του συστήματος, αλλά και στον προγραμματιστή του λογισμικού, διότι περί αυτού πρόκειται, για το λογισμικό εδώ. Και στην προκειμένη περίπτωση, ίσως από πολιτικής πλευράς, να μην επιθυμεί κάποιος να έχει την ευθύνη ο χρήστης ε, ε, αυτή τη στιγμή που άρχει αυτόνομη οδήγηση βέβαια, ο χρήστης ε, πάντοτε είναι αυτός, αλλά ίσως να μην δίνεται το σωστό μήνυμα. Δεν είναι σωστός πως διότι ο, ο χρήστης ναι μεν χρησιμοποιεί το όχημα, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει, άρα δεν μπορεί να κάνει καμία αλλαγή αν δούμε επικοινωνία μηχανήματος προς μηχάνημα, εκεί ίσως ο κατασκευαστής που χρησιμοποιεί το μηχάνημα θα μπορούσε να έχει και την ευθύνη μπορεί να είναι ε, τώρα ε, στο νέο σύστημα αυτός ο υπεύθυνο. Ε, θα έλεγα όχι γιατί υπάρχει ένας περιορισμός εδώ με το λογισμικό για παράδειγμα. Ο προγραμματιστής τώρα του λογισμικού δεν ωφελείται τελικά, δεν έχει το όφελος από το προϊόν που πηγαίνει εκεί το λογισμικό. Άρα ούτε και εδώ θα μπορούσαμε επομένω να θεωρήσουμε ότι υπεύθυνο είναι ο κατασκευαστής του συστήματος που στην τσέπη του πηγαίνει το κέρδος. Και βέβαια πρέπει να το συνδυάσουμε και με την ασφάλεια. Γιατί το σύστημα ναι μεν είναι αυτόνομο, αλλά τι θα γίνει αν δεν λειτουργεί σωστά και δεν υπάρχει αμέλεια. Τι γίνεται εκεί. Πρέπει να βρεθεί μια προσπάθεια με την ασφάλεια, με την ασφάλιση. Άρα νομίζω πρέπει να εστιάσουμε στον κατασκευαστή που ασχολείται με το όλο σύστημα, το ρομπότ, αυτό, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει και εκεί συνδεδεμένη ε, η ευθύνη. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε επιπλέον ένα λεγόμενο e-person, δηλαδή κάθε ρομπότ, κάθε σύστημα να έχει νομική προσωπικότητα. Η απάντηση είναι όχι, η δική μου απάντηση, διότι δύο πράγματα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρώτον, την ευθύνη και εδώ πρέπει να αποδοθεί κάπου πίσω από το ρομπότ, σε, κάποιον, σε κάποιο πρόσωπο. Δεν χρειάζεται αυτό το e-person ως κάτι προσωρινό ή ενδιάμεσο. Μπορεί να αποδοθεί ευθύνη στον κατασκευαστή ή να συνδυαστεί με την λύση της ασφάλειας, της ασφάλισης. Άλλη επιλογή. Και γιατί είμαι κατά του να έχω αυτό το e-person. Αν αυτό παραγγέλει ή ε, τιμολογεί ή αποφασίζει ποιο προϊόν θα αγοραστεί. Αν γίνει αυτό, τότε αυτό το πρόσωπο θα πρέπει να είναι μια τεχνητή νομική οντότητα, τεχνητό νομικό πρόσωπο που θα το αποδοθεί αυτή η ευθύνη. Εγώ απαντώ και εδώ αρνητικά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πάντα πρέπει αυτό το ρομπότ να το συνδυάσουμε, να το συνδέσουμε με το κατασκευαστή που το χρειάζεται αυτό το υλικό που έχει παραγγείλει το άλλο πρόσωπο. Και πάντα αυτή η δήλωση του e-person θα πρέπει να συνδέεται με τον κατασκευαστή που το χρειάζεται. Και εκεί έχουμε τις διορθώσεις βαλμάτων κτλ. και Τα συνήθη. Big data, μαζικά δεδομένα, μείζον θέμα πρέπει να συζητήσουμε. Υπάρχουν δύο συζητήσεις που γίνονται εκ παραλίλου. Ε, η πρώτη είναι ο νόμος θα πρέπει να διέπει την ιδιοκτησία των δεδομένων, δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, για την παραγωγή για παράδειγμα, από το εργοστάσιο. Και το δεύτερο είναι ο ιδιωτικός χαρακτήρας των δεδομένων. Χρειάζεται ένα είδος κανονισμού για την πρόσβαση στα δεδομένα, ένα είδος κυριότητας ιδιοκτησίας δεδομένων. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν διάφορες απόψεις και σκέψεις. Θα πρέπει να δούμε και την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και το πώς θα ορίζαμε αυτά του, αυτού του είδους τα δεδομένα. Και από εκεί και πέρα η υφιστάμενη νομοθεσία αρκεί ή όχι. Ας έρθουμε τώρα σε αυτό το θέμα και να το δούμε σε βάθος. Για τα προσωπικά δεδομένα έχουμε την νομοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ το 2018, όπου ρυθμίζεται ξεκάθαρα το τι είναι προσωπικό δεδομένο, τι δεν είναι όμως, τι είναι το non-personal data, σας πω εγώ, 11 βαθμοί Κελσίου. Αυτό τι είναι, μη προσωπικό δεδομένο, αλλά σας ε, χρησιμεύει η πληροφορία το ότι είναι 11 βαθμοί Κελσίου ή μόνο αν σας πω ότι είναι 11 ε, βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία του μηχανήματος ή ε, έξω η εξωτερική θερμοκρασία, άρα είναι πολύ κρύα ατμόσφαιρα για το μηχάνημα. Μόνο λοιπόν αν υπάρχει ένα συνδυασμό αυτών των πληροφοριών έχει νόημα. Πώ ορίζουμε όμω τελικά τι την χάνει προστασία ε, μέσω τη νομοθεσία. Θα μπορούσε κανεί να εστιάσει μόνο στον, κωδικό, στον κώδικα. Δι, είναι διαδικό, παραδείγματο χάρη, binary code και τα προστατεύουμε όλα, αλλά υπάρχουν προβλήματα εκεί. Γιατί αν προστατεύουμε τα πάντα θα χρειάζεται να προστατεύουμε και τι πληροφορίε και εκ παραλλήλου να ρυθμίσουμε και να νομοθετήσουμε και για την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. επομένω. το ισχύον δίκαιο, η ισχύουσα νομοθεσία, θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι μια χαρά. Έχουμε ε, για τι αθέμητε πρακτικέ νομοθεσία, για την προστασία εμπορικού απορρίτου, επιχειρηματικού απορρίτου, για τα προσωπικά δεδομένα κτλ. κτλ. Και έχουμε και το database law που έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ευρώπη είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Να μπορούσαμε ίσως ε, να το βρούμε πολύ χρήσιμο. Χρειάζεται λοιπόν νέα νομοθεσία. Και για ποιο λόγο για να προστατεύσουμε την καινοτομία. Γιατί, μα δεν υπάρχει καινοτομία, γιατί εδώ μιλάμε για συλλογή δεδομένων. Δεν υπάρχει δημιουργική πράξη από πίσω. Το χρειαζόμαστε αυτό μήπω για τη διαφάνεια των αγορών, για την ψηφιακή αγορά. Χρειαζόμαστε ένα νέο κανονισμό. Μέχρι στιγμή δεν έχω διαπιστώσει να υπάρχει κάποια στοχεία τη αγορά. Γιατί λοιπόν να κάνουμε μια νέα ρύθμιση ή μήπω θέλουμε να εξισορροπήσουμε κάποια κενά ε, ισχύω εξουσία. Αλλά αυτό πάντοτε υπάρχει. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μια νομοθεσία εδώ η οποία είναι στο πλαίσιο του ενοχικού δικαίου. Έχουμε τα περί προστασίας δεδομένων. Και τώρα σε ό,τι αφορά την, τον ιδιωτικό χαρακτήρα των δεδομένων, έχουμε κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Privacy by Design, έχουμε την ανωνυμοποίηση και ψευδοανωνυμοποίηση, Άρα δεν χρειαζόμαστε εδώ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και αν χρειαζόμαστε τέτοιου είδου δεδομένα έχουμε ένα τεράστιο εμπόδιο λόγω τη αρχή ε, του ε, ειδικού σκοπού. Πρέπει να προσδιοριστεί ο σκοπό. Αν χρειαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ή μαζικά δεδομένα στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί υπάρχει αυτή η αρχή. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εσείς θέσετε πολύ σημαντικά ερωτήματα για τα αυτόνομα συστήματα, ποιος φέρει την αστική ευθύνη για τα προϊόντα, τι είστε ηλεκτρονικό πρόσωπο, ποιο συνδέεται με τα big data και μαζικά δεδομένα και ποιο τα χρησιμοποιεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σα. Επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Έντι Ρούλαντς, αντιπρόεδρο της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας στην εταιρεία Siemens. ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του πριν από λίγα χρόνια στη Siemens. Ε, όχι και τόσο λίγα. Ναι, ήταν ακόμα 20ος αιώνας, λέει ο πρόεδρος, όταν αρχίσατε. Έχετε σπουδάσει οργανική χημεία και έχετε και διδακτορικό. Ε, και εργάζεστε στη Siemens στα γραφεία των Βρυξελών από το 2004. Ε, είναι πολύ σημαντική η έρευνα, η καινοτομία, αλλά καθώς επίσης και τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, πάρα πολύ σημαντικά φυσικά και ε, επίκαιρα θέματα και ενδιαφέροντα για μας. Έχετε μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη που είχατε να με καλέσετε. Σήμερα θα επικεντρωθώ στην ψηφιοποίηση της παραγωγής ε, δηλαδή ε, βιομηχανία 4.0 η λέξη κλειδί. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ψηφιοποίηση άρχισε από τους καταναλωτές, ας πούμε από τα βιβλία, πήγαμε σε ηλεκτρονικά βιβλία, από ε, τα CD περάσαμε σε streaming και τώρα έχουμε περάσει και από επιχείρηση σε επιχείρηση, business to business. Και βλέπετε εδώ τους διάφορους τομείς που καλύπτει η Siemens, αλλά εμείς θα ασχοληθούμε με την ψηφιοποίηση 4.0, με την ψηφιακή παραγωγή. Η ίδια ψηφιοποίηση είναι ε, δημιουργία της αρχής, από την αρχή μάλλον από τη σύλληψη και το σχεδιασμό του προϊόντος μέχρι το τέλος που μιλάμε για τη συντήρηση και για την επισκευή. Και αυτό ισχύει για όλους αυτούς τους κάθετους τομείς που βλέπετε στην παρούσα διαφάνεια. Πάντα υπάρχουν ε, κινητήριες δυνάμεις και προκλήσεις, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σήμερα είναι πολύ πιο περίπλοκα τα προϊόντα, όπως είπε και ο συνάδελφος από το Fraunhofer, ε, ο καταναλωτής θέλει πιο εξατομικευμένα προϊόντα. Έχουμε μαζική παραγωγή αλλά με χαρακτηριστικά προσωπικά. Ε, χάνουμε δεδομένα αλλά αυξάνουμε την ποιότητα Παλλον χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προς ε, την κατεύθυνση αυτή και η οικονομία ενέργειας ε, γενικά είναι πολύ σημαντική. Ε, το Industry Platform 4.0 είναι ένα γερμανικό σχέδιο που στοχεύει στη βιομηχανική παραγωγή μετά το έτος 2025 και στόχο έχει προσπαθεί τουλάχιστον να λύσει όλες αυτές τις νέες προκλήσεις και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την ψηφιοποίηση της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Δηλαδή τι κάνει, συμπεριλαμβάνει όλες τις από την ίδια την ιδέα της σύλληψη του προϊόντος μέχρι την παραγγελία και όλες τις ε, υπηρεσίες μετά την πώληση. Ε, το ονομάζουμε Digital Twin αυτό, ένα ψηφιακό δίδυμο, το ανέφερε προηγουμένως συνάδελφος από το Fraunhofer. Βλέπετε εδώ τις φωτογραφίες ε, στη διαφάνεια κάτω που είναι η πραγματική γραμμή παραγωγής και η αλυσίδα παραγωγής αξίας. Εκεί έχετε μια τελείως ψηφιακή μορφή ε, στην ε, διαδικασία της παραγωγής, αλλά πριν την παραγωγή υπάρχει ο σχεδιασμός, ε, η κατασκευή, η παραγωγή του προϊόντος κτλ. Υπάρχει και η βιομηχανία που, χρησιμοποιεί κάποιες μεθόδους που δεν παράγει προϊόντα, αλλά είναι αντίστοιχη αυτή και η ψηφιοποίηση και τελικά σε ένα εργοστάσιο χημικό, ας πούμε. Εδώ δεξιά βλέπετε πάλι μια διαφάνεια για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει ένας παραλληλισμός του εικονικού με τον πραγματικό κόσμο και πώς μεταφέρεται εδώ όλα τα δεδομένα που παράγονται σε όλη τη διαδικασία της πραγματικής γραμμής παραγωγής μπορούν να χρησιμοποιούνται κάθε φορά για να βελτιώνεται η προηγούμενη φάση της μεθόδου και η επόμενη. Ποια είναι τα τέσσερα βασικά ε, συστατικά τα βλέπετε εδώ αριστερά. Πρώτον, χρειάζεται ένα βιομηχανικό λογισμικό και ένα χαρτοφυλάκι αυτοματοποίηση. Αυτό το ονομάζουμε εμεί ψηφιακή εταιρεία, που θα πρέπει κάθε φορά να το σχεδιάσετε για τους πελάτες σας, ε, όταν δεν παράγεται ε, προϊόντα συγκεκριμένα, αλλά μεθόδους. Δεύτερον, ε, βιομηχανική επικοινωνία, δίκτυα επικοινωνία, βεβαίω προστατευόμενη ε, για να προστατεύετε και η πνευματική σας ιδιοκτησία. Υπάρχει και θέμα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και στη βιομηχανία. Ε, και τέλος έχουμε τις βιομηχανικές υπηρεσίες για τους πελάτες. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ε, μέσων που ονομάζονται κοινέ πλατφόρμες για αυτό το είδος της βιομηχανίας. Έρχομαι σε ένα παράδειγμα τώρα πολύ ουσιαστικό από την πράξη. Η παραγωγή μαζεράτη τώρα ε, ε, γίνεται απολύτως με αυτό τον τρόπο με την ψηφιακή μορφή. Και παράλληλα χρησιμοποιούνται και εικονικά και πραγματικά δεδομένα για να βελτιστοποιείται η παραγωγή στο σύνολό της από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι το τελικό προϊόν. Για να, ε, και έχει αυξηθεί κατά 30% η αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, ο χρόνος ε, μέχρι να φτάσει στην αγορά που ήταν 4 χρόνια από την παραγγελία, τώρα έχει φτάσει στους 32 μήνες με τον τρόπο με τον οποίο σήμερα εργαζόμαστε. Είναι ε, λόγος για ρομπότ. Βλέπετε εδώ ένα φιλμάκι για το πώς παράγεται ένα αυτοκίνητο σήμερα. Παίρνουν τα στοιχεία τα ρομπότ, συζητούν μεταξύ τους, περιμένουν το ένα το άλλο να κάνει τη δουλειά του ε, συναρμολογούν το αυτοκίνητο και μετά προχωράει στο επόμενο βήμα. Ε, δηλαδή όλες οι μεταβλητές που υπάρχουν σε ένα τέτοιο ε, εργοστάσιο περνάνε μέσα από τα ρομπότ. Είναι και διαφορετικές και διαφορετικά προγράμματα και θα πρέπει όλα αυτά να προγραμματίζονται. Αύριο όμως τι θα γίνει όταν μιλάμε για τελείως αυτόνομα συστήματα και πιο ευφυή συστήματα. Οι αυτόνομες μηχανές δηλαδή ήδη μπορούν ανεξάρτητα να κοιτάξουν τι χρειάζεται και τι τύπος είναι ε, το αυτοκίνητο <laughs> αυτό που πρέπει να κατασκευαστεί. Τους δίνουμε μια συνταγή με τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που περιμένουμε να το κάνουν, αλλά δεν τα προγραμματίζουμε, αποφασίζουν μόνα τους τον τρόπο με τον οποίο θα έχουν, ε, δημιουργούν ε, κώδικες παραγωγής ε, και κατασκευάζουν ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου ή του οχήματο που χρειάζεται. Βεβαίω και ε, οι άνθρωποι συνεργάζονται ακόμα με τι αυτόνομε μηχανέ πολύ στενά και είναι και ανάγκη να αναγνωρίζουν τα ρομπότ ε, τον άνθρωπο, ότι υπάρχει δίπλα τους ένας άνθρωπος και να προσέχουν ε, με ποιο τρόπο δουλεύουν και να επιταχύνουν όταν δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί γύρω που να κινδυνεύει να τον χτυπήσουν. Τώρα, ε, τα μεγάλα μαζικά δεδομένα και τα εφή δεδομένα. Βλέπουμε εδώ τα προϊόντα της Siemens. Έχουμε 300.000 περίπου συσκευές παγκοσμίως ε, της Siemens ε, που ε, είναι εγκατεστημένες και μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι τομογράφος, ιατρική συσκευή, συσκευή παραγωγής ενέργειας, τουρμπίνες, τα λοιπά ε, Παράγουν δεδομένα. Για να τα αναλύσουμε θα πρέπει να έχουμε μια γνώση για το κάθε χώρο. Δηλαδή είναι από την υγεία, είναι από την ενέργεια, είναι από τις μεταφορές. Θα πρέπει να γνωρίζουμε το πλαίσιο, ε, την τεχνογνωσία και να έχουμε κάποια ιδέα χονδρικά για ε, την αναλυτική και τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούν. Και μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία για να βγάλουμε τα ευφύ δεδομένα που βοηθάνε και εμάς και κυρίως τους πελάτες για να αυξήσουν την παραγωγή τους με μείωση του κόστους, με εξοικονόμηση ενέργειας όπως σας είπα. Και ένα καλό παράδειγμα γι' αυτό είναι φυσικά αυτό που θα γνωρίζετε στο ΣΕΡΝ, αυτό το μεγάλο επιταχυντή σωματιδίων που παράγει και στοιχειώδη ε, θεμελιώδη σωματίδια. Είναι 27 ε, ε, χιλιόμετρα, ε, ε μείον 291 βαθμούς Κελσίου, έχει ε, ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου για 600 ελέγχους, συν 18.000 αισθητήρε και όλα αυτά τα δεδομένα τα χρησιμοποιεί η Siemens για να τσεκάρει το σύστημα, να κάνει ένα ε, check-up για να δει αν υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας. Δεν μιλάω καθόλου για τα επιστημονικά δεδομένα που παράγονται, μόνο για τα δεδομένα λειτουργίας. Για να ε, μπορεί να λειτουργεί αυτή η μηχανή και να αυξάνει ε, τη λειτουργία τους. Τη μέρα έχουμε 100 terabytes δεδομένα, ένα 24ωρο. Ταυτόχρονα αυτό το μηχάνημα κάθε ε, ε, δευτερόλεπτο ε, παράγει περίπου 40 τεραμπάιτ δεδομένων επιστημονικών. Όλα αυτά λοιπόν γίνεται με την αναλυτική που επιτρέπει να βελτιωθεί η μηχανή αυτή. Στο παρελθόν χρειαζότανε 14 μέρες, δύο εβδομάδες για να βρεις που είναι το λάθος τα 27 χιλιόμετρα, ενώ τώρα χρειαζόμαστε περίπου μισή ώρα για να δούμε που υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα και μαζικά δεδομένα και ευφύ δεδομένα. Τελειώνω με αυτή τη διαφάνεια που σας δείχνω εδώ, όπου δεξιά βλέπετε το ε, ε, Internet of Things, ε, το διαδίκτυο των αντικειμένων για τους πελάτες μας που έχουν εργοστάσια, κρίσιμες υποδομές, μπορεί να είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας ή κάτι από την ιατρική ή στο ΣΕΡΝ, έχουν ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αστική ευθύνη, με το σέρβις, με την προστασία των δεδομένων. Εμείς το αφήνουμε στα χέρια του πελάτη. Όλα τα, τα, τα στοιχεία, τα δεδομένα τα στέλνει στο cloud και τα ε, ελέγχει αυτό ή φέρνουμε έναν υπολογιστή πολύ κοντά στο μηχάνημα έτσι ώστε ήδη να δημιουργούνται εκεί, να παράγονται ευφύ δεδομένα και να αποστέλλονται σε εμά, ας πούμε στη Siemens όπου χρειάζεται συντήρηση, όπου χρειάζεται service. Αλλά τα ίδια τα δεδομένα, τα βασικά του, του, του κατόχου ε, του μηχανήματος δεν φεύγουν από αυτό. Αυτό το λέμε το web των συστημάτων, γιατί τα συστήματα επικοινωνούν μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να περάσουμε πάντα από το διαδίκτυο με τα δεδομένα. Αυτό είναι κάπως διαφορετική φιλοσοφία που είναι προσανατολισμένη στον πελάτη, ε, στον τομέα business to business από επιχείρηση σε επιχείρηση. Νομίζω ότι τελείωσε η ώρα μου. Ε, ξεπέρασα κατά 20 δεύτερα. Να με συμπαθάτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, τώρα θα μιλήσουμε για ένα νέο σύστημα για τη ρομποτική, αυτοματοποιημένα συστήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Enterprise. Νομίζω θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη μελλοντική νομοθεσία. Ο κύριος Κεκαλάινεν είναι ο τέταρτος ομιλητής, εκτελεστικός διευθυντής της ΕΝΕΒΟ εσείς είσαστε ένας ε, πολύ σοβαρός επιχειρηματίας, είσαστε ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΝΕΒΟ, που είναι μια φιλανδική νεοσύστατη εταιρεία που ασχολείται με την διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωσή τους. Και αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να βρείτε έναν οικονομικό τρόπο περισυλλογής αποβλήτων για τις ε, μεγάλες πόλεις. Έχετε το λόγο. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ. Εγώ είμαι ένας επιχειρηματίας, ε, δεν είμαι ούτε καθηγητής ούτε δόκτωρ και θα σας δώσω ένα έμπρακτο παράδειγμα για το πώς ε, μπορούμε να συλλέξουμε δεδομένα για την διαχείριση μιας πολύ παραδοσιακής αλλά ευρύτατης ε, βιομηχανίας. Τώρα για την εταιρεία μου. Το 2010 συστάθηκε η εταιρεία και χρησιμοποιούσαμε από κατεφροτές ε, για την ε, όλη διαδικασία διαχείρισης, αλλά στη συνέχεια είδαμε ότι η βιομηχανία των αποβλήτων μπορούσε να αλλάξει χρησιμοποιώντας ε, την τεχνολογία για να δούμε τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά. Η έδρα μας είναι στη Φιλανδία, από όπου κατάγομαι και εγώ. Έχουμε ανοίξει πολλά γραφεία και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία. Ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά η διαχείριση, η παγκόσμια διαχείριση αποβλήτων είναι μια τεράστια βιομηχανία. Είναι πολύ μεγαλύτερη από την κινητή τηλεφωνία κάτι που δεν θα το φανταζόμασταν. Πρόκειται για μια αγορά ενός 3 ε, ε, ευρώ και αυξάνεται ετησίως λόγω των ε, μετατάσεων της οργάνωσης και λοιπά, διαχείρισης και λοιπά. Όσοι ζουν ε, σε αστικές περιοχές παράγουν δύο φορές ε, παραπάνω απόβλητα από, τις, από εκείνους που κατοικούν στις αγροτικές περιοχές. Υπάρχουν εκατοντάδες ε, κοντέινερ απορριμμάτων και εκατομμύρια φορτηγά που τα περισυλλέγουν. Μιλάμε για ένα Το όμως, το 50% με συγχωρείτε, είναι η η μελητιακή υποστήριξη. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο έχουμε πραγματικά δεδομένα και δεν κάνουμε εικασίες. Έτσι έχει η κατάσταση. Έχουμε απορριμματοφόρα που μεταφέρονται από το ένα σημείο στο δεύτερο σημείο για να μεταφέρουν ε, απόβλητα. Πρόκειται για μία διαδικασία μετακίνησης και δεν ξέρουμε πόσα απόβλητα παράγονται κάποια τη, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θέλουμε όμως αυτό το στατικό μοντέλο να γίνει δυναμικό, να ξέρουμε πού να πάμε, πώς, ποια χρονική στιγμή ανάλογα με την ε, ε, με τα απορρίμματα που δημιουργούνται. Αυτή την εικόνα την ξέρετε. Η μία είναι από τη Φιλανδία, αυτή είναι από τη Φιλανδία, πριν είδατε μία εικόνα από τη Βαρκελόνη. Αυτό είναι πρόβλημα. Πολλές φορές αργούμε πάρα πολύ στην ε, περισυλλογή των αποβλήτων και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε αυτούς τους αισθητήρε και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι πότε, σε πόσο χρονικό διάστημα ένα φορτηγό γεμίζει από, ε, απορρίμματα, απόβλητα για να ξέρουμε και πότε πρέπει να αδειάσουν και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε τις διαδρομές μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ σωστό στόλο έχουμε μειώσει το κόστος κατά 50% από πλευράς επιμελητίας και αυτό σημαίνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Οι αισθητήρε είναι ε, μία μέθοδος για να συλλέγουμε πληροφορίες. Συλλέγουμε πληροφορίες, ξέρουμε πως έχει θερμοκρασία, ε, τι κίνηση υπάρχει και τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε κοντέινερ. Τα ευεργετήματα είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε χαμηλότερο κόστος και αν ξέρουμε πόσα απόβλητα δημιουργούνται, παράγονται, τότε ξέρουμε πώς μπορούμε και να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί υπάρχουν πολλές επιπτώσεις και στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, ως προς μέταλλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 75% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με οποιαδήποτε άλλα υλικά. Ε, εδώ μιλάω για πρώτες ύλες και πώς μπορούμε να τις ανακυκλώσουμε καλύτερα. Άρα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και νέα ε, συστήματα δεν χρειάζεται να πάμε πίσω στις πρώτες ύλες. Εδώ είναι μερικοί από τους πελάτες μας στην Ευρώπη. Η Ολλανδία είναι στην εμπροστοφυλακή της ε, περισυλλογής. Η Ισπανία, οι βόρειες χώρες, πολλές ε, χώρες της Βόρειας Ευρώπης, το Λονδίνο και η περιφέρειά του ε, εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε και με τη Νέα Υόρκη βλέπουμε ότι αλλάζουν οι τεχνολογίες και αλλάζει και ο τρόπος διαχείρισης. Η τεχνολογία βοηθάει σε αυτές τις αλλαγές. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία όσο περισσότερο μπορούμε για να γίνουν όλα πιο αποδοτικά και να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες. Επίσης, στην Ιαπωνία μας ήταν πολύ επιτυχημένη και είναι πολύ περίεργο για μια νεοσύστατη εταιρεία της Ευρώπης να επικρατεί στην Ιαπωνία. Και αυτό δείχνει πόσο πραγματικά έχουμε προοδεύσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Είναι ένα πολύ απτό παράδειγμα για το πώς λειτουργούν τα πάντα. Μιλάμε, μιλήσατε για τη σημασία της διαχείρισης αποβλήτων σε σχέση με την κινητή τηλεφωνία, το εμπλεκόμενο, το ενεχόμενο κόστος. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στις ερωταποκρίσεις. Ο κύριος Μπόνι από πλευράς του ΕΛΚ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις που μας ενέπνευσαν. Το ίδιο και οι απόψεις για τη βιομηχανία 4.0 και για τα ρομπότ και τα μαζικά δεδομένα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας για να αποκτήσουμε ως Ευρωπαϊκή Βιομηχανία ένα νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Έχω έτσι κάποια σημεία για να δώσω τροφή στη συζήτηση. Καταρχάς, οι συνθήκες ε, για την ανάπτυξη του τομέα αυτού, η συνδεσιμότητα, τι άποψη έχετε για όλα αυτά, ενώ υποδομές υψηλής ποιότητας υποδομές και δίκτυα κέντρα υπολογιστών υψηλών επιδόσεων και στην Ευρώπη εν γέννη. Επίσης, επικοινωνία μεταξύ όχι μόνο των χρηστών ως ανθρώπων, αλλά και η επικοινωνία μεταξύ των μηχανημάτων που μπορεί και αυτά να είναι χρήστες. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερες υποδομές για την ανάπτυξη αυτού του τομέα. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να αναφέρω, ο κύριος Πούτς το ανέφερε, δεδομένα ως πηγή. Συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα της ιδιοκτησίας, της κυριότητας των δεδομένων. Ποιο είναι αυτό όμω που παράγει τα δεδομένα για τις αυτές τις διεργασίε. Τα δεδομένα παράγονται όχι μόνο από ανθρώπους, αλλά πολλές φορές παράγονται αυτόματα από μηχανές. Άρα οι κανόνες είναι σημαντικοί για την προστασία των δεδομένων, την ασφάλεια των δεδομένων. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια διάκριση άλλο τα προσωπικά δεδομένα και άλλο αυτά παράγονται από μηχανήματα. Και πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της κυριότητας των δεδομένων και πώς πρέπει να θέσουμε και το πρόβλημα της συνειδητοποίησης ότι η οικονομία αυτή βασίζεται στην επεξεργασία δεδομένων πρώτα απ' όλα. Τρίτος τομέας. Οι νέες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ. Συμφωνώ ότι χρειάζεται κανόνες συνεργασίας. Και χρειάζεται και καλύτερη επικοινωνία. Και αν κατάλαβα καλά, δεν μιλάμε μόνο για συνεργασία μηχανική, αλλά μιλάμε και για την χρήση της δικής μας της φωνής ως ανθρώπων. Υπάρχουν τώρα κάποιες φωνητικές εφαρμογές. Είναι σημαντικό η φωνή μας, για παράδειγμα, μέσω των ε, φιών ε, τηλεφών, των smartphone, να ε, στέλνεται στα μηχανήματα. Τι επικοινωνία λοιπόν χρειάζεται όταν θα συνεργαστούμε με τα ρομπότ εμείς οι άνθρωποι και πώς περιγράφεται αυτή η ευθύνη, τα πολύ ενδιαφέρουσα η έννοια που μας παρουσίασε ο καθηγητής Μπρόιτιγκαν για το, για το ηλεκτρονικό πρόσωπο e-person. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για κάποιες ευθύνε ε, με την παραδοσιακή έννοια του όρου, γιατί εδώ χρειαζόμαστε εντελώ νέες λύσεις. Και πρέπει να τις σκεφτούμε. Να πω επίσης ότι η Επιτροπή Γιούρη έχει ξεκινήσει εργασίες στις οποίες πιστεύω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Τέλος, συμφωνώ ότι χρειάζονται κανόνες, αλλά δεν πρέπει και να το παρακάνουμε, να έχουμε τελικά υπερρύθμιση. Τέλος, τυποποίηση. Μας δίνει η ψηφιακή τεχνολογία πολλές νέες δυνατότητες για τη μελέτη και σχεδιασμό προϊόντων αλλά και υπηρεσιών και για τυποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα και εξατομήκευση υπηρεσιών προϊόντων. Αυτό παρέχει προσθέμενη αξία και είναι ένα πλεονέκτημα αυτού του κλάδου βιομηχανία 4.0. Όμως, όπως ανέφερε και ο κύριος Ρόλαντς, κοινέ πλατφόρμες, δηλαδή βιομηχανική επικοινωνία, ασφάλεια και υπηρεσίες από κοινού. Πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν τις πλατφόρμες ε, με έναν νέο τρόπο. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί ήταν πολύ αποδοτική. Ναι, αλλά μακρηγορείτε, λέει ο πρώτος, μακρηγορείτε. Mm. Ναι. Τέλος πάντων, ο κύριος Μπον, ένα τελευταίο, τελευταίο, για τη ρύθμιση. Ε, Το και... θα έχουμε χρόνο ε, για μετά. Ε, κύριε Βεν, από σοσιαλιστές και δημοκράτες. Συγγνώμη σας διέκοψα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μιλήσαμε πάρα πολύ τώρα για τα τεχνολογικά ζητήματα της βιομηχανίας 4.0, για θέματα ε, εταιριών, κατασκευαστριών, ε, δράση, νέα μοντέλα, επιχειρηματικά, νέες νοοτροπίες. Εγώ θα ήθελα να φερθώ σε ένα διαφορετικό στοιχείο, το εξής ε, αυτό το θέμα δεν θα πρέπει να απασχολεί μόνο τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών για να βρουν νέα επιχειρησιακά μοντέλα και νέα ρίσκα. Οι εργαζόμενοι τι γίνεται, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την ε, προσπάθεια ε, άνδρες και γυναίκες. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν από τη δική σας εμπειρία σε ποιες εταιρείε αυτό ε, λειτουργήσε ιδιαίτερα καλά, ή αν υπάρχουν και ε, κλάδοι ε, τι γίνεται με την κατάρτιση, τη μετακπαίδευση, τη συμπερίληψη των επιχειρησιακών συμβουλίων, ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων, μελέτες, πώς συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σε αυτή την προσπάθεια εμεις μήπως χρειάζονται νέες μελέτες για το πώς το βλέπουν οι εργαζόμενοι. Γενικά κάπως αυτό μου φάνηκε ότι έχει παραγωνιστεί στη συζήτηση. Ε, βλέπετε την ανάγκη ενδεχομένω κοινωνικού διαλόγου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερη ερώτηση. Εδώ στην Επιτροπή μα μας απασχολεί ε, και το θέμα τη αστική ευθύνη ε, των ρομπότ. Πολύ ωραία τα αναφέρατε αυτά εσείς κύριε Μπρόιτιγκαν και σε σχέση με τα μαζικά δεδομένα. Έχω μια ερώτηση που θα έχουν και άλλοι συνάδελφοι και τον έφερε προηγουμένως με τις υποδομές. Τι χρειαζόμαστε για να διευρυνθεί η ευρυζωνικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου, ο Πρόεδρος. Ο, ο κύριος Τοσινόφσκι από τους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Κατά την άποψή μου είναι και πάρα πολύ επίκαιρα. Σήμερα στο Κοινοβούλιο σε διάφορες επιτροπές συζητούμε ε, τι θέση πρέπει να έχουν τα ρομπότ στη ζωή μας. Ε, πώς αναπτύσσονται, πώς γίνεται η έρευνα, ε, πώς δηλαδή από εδώ και πέρα ε, θα έχουμε ε, μεθόδους τυποποίησης ε, έτσι ώστε να υπάρχει και ένα είδος φρένου, να έχουμε μια τροχοπέδη για να μπορούμε να ελέγχουμε και τα ρομπότ. Θέλω λοιπόν να σας κάνω την εξής ερώτηση. Ο νομοθέτης προς τα που θα πρέπει να κινείται. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Μπρόιτιγκαμ. Είπε ότι δεν θέλω να επαναλάβω επιλέξει αυτά που είπατε, αλλά είπατε ότι η σημερινή νομοθεσία αρκεί. Δεν χρειάζεται νέα νομοθεσία. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό ισχύει. Ε, πολύ συχνά ε, νομοθεσία που διέπει την έρευνα και ανάπτυξη δεν είναι πάντα προς όφελός της, μπορεί να τη φρενάρει κιόλας. Ερωτώ λοιπόν και σας λέω την άποψή μου μήπως θα πρέπει να κινηθούμε περισσότερο προς την εκπαίδευση, την παιδεία, τις υποδομές, την κατάρτιση ε, για να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Ε, ε, ευρυζωνικότητα, τεχνολογίες πληροφορικής κτλ. Γιατί φοβάμαι ότι αν το παρακάνουμε στην νομοθεσία θα στραγγαλίσουμε ε, και θα φρενάρουμε τις εξελίξεις. Και η τεχνολογία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς ε, που δεν μπορεί πάντα να ακολουθεί μια διοίκηση και μια νομοθεσία. Η τεχνολογία ε, μας ξεπερνάει, ακολουθεί τους δικούς τους νόμους, δεν, δικούς τους νόμους, δεν περιμένει τους νόμους των κρατών. Θα ήθελα λοιπόν να πω ε, κάτι σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Ρούλαντς. Αν είμαστε υπερβολικά ε, παρεμβατικοί και χρησιμοποιούμε αυτές τις μεθόδους υπερβολικά, ε, μπορεί αυτό να είναι πρόβλημα. Και θα έχουμε τελικά ένα μοντέλο αυτοκινήτου. Γιατί τα ρομπότ θα βγάζουν πάντα τον ίδιο τύπο αυτοκινήτου. δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό. Σας ερωτώ λοιπόν, το Κοινοβούλιο τι λέτε ότι πρέπει να κάνει, πού βλέπετε το ρόλο του και πώς τον θεωρείτε. Eh, θα πρέπει να είμαστε ακτιβιστές ή ε, να έχουμε άλλη προσέγγιση διαφορετική. Να ξεπεράσουμε τους φραγμούς και τις παραδοσιακές ε, νοοτροπίες. Για να προλάβουμε ε, αυτή την ανία και την ομοιομορφία. Εγώ θέλω να έχω διαλέγω μοντέλο, όχι ένα ενίο μοντέλο αυτοκινήτου. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το τελευταίο. Τι ρωτήσατε όμως ακριβώς, ότι πώς θα έχουμε βιομηχανική δραστηριότητα χωρίς παρέμβαση ανθρώπων και χωρίς παρέμβαση Κανενός Θεός φυλάξει. Καλά, θα δούμε λοιπόν. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Ο συνάδελφος Beauty από τους Πρασίνους. Thank you, Chair. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριοι για τις παρουσιάσεις αυτές. Έχω ορισμένε ερωτήσεις προς τον κύριο Πούτς. Είπατε, εν ότι και η Κίνα ασχολείται με την ε, πρόθεση αυτής της τεχνολογίας, αυτού του τεχνολογικού άλματος. δηλαδή έχουν ορίσει την στρατηγική Made in China 2025 σε σχέση με τους απότερους στόχους της χώρας. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι, ποιες είναι οι δικές σας συμβουλές για το ποια στρατηγική θα πρέπει να ακολουθήσουμε ως Ευρώπη, γιατί γνωρίζετε την υπόθεση Κούκα και ο Επίτροπος Έτιγκερ εξέφρασε την απόψή του και είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να υπερασπιστεί τη βιομηχανία, τις βιομηχανίες και τεχνολογίες στρατηγικής σημασίας εάν θέλει να είναι στην πρωτοπορία, να παραμείνει στην πρωτοπορία. Υπάρχουν ανησυχίες σε σχέση με την Κίνα επί του θέματος. Δεύτερον, δεν μας μιλήσατε για τις ε, ΜΜΕ, κυρί. Μιλάμε για μία διαδικασία τυποποίησης αυτών των νέων τεχνολογιών από τις ΜΜΕ. Και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο μας συμβουλεύετε να ακολουθήσουμε την τυποποίηση από ευρωπαϊκής κοπιάς και διεθνούς κοπιάς τι μας προτείνετε. Και σε σχέση με τις ψηφιακές δεξιότητες, είναι ευρέως γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού μας δεν έχει τις ε, κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες. Θα είχε νόημα μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση από τη πλευρά της ανάπτυξης μιας ενίας ψηφιακής αγοράς θα είχε νόημα κάτι τέτοιο. Αλλά αν μιλήσουμε για αρμοδιότητες, εδώ έχουμε να κάνουμε με τα κράτη-μέλη ή και με περιφερειακές αρμοδιότητες ακόμα. Πώς να το διαχειριστούμε. Ο κύριος Κόχλιτσεκ, ο αντιπρόεδρος μας από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα μιλήσω τσεχικά όπως και ο ε, προλαλής σας ε, συμπατριώτης μου. Έχουμε δίκτυα ευρυζωνικά. Δηλαδή είμαστε σε θέση τα δεδομένα να τα μεταφέρουμε σχετικά γρήγορα. Ωραίο είναι αυτό και καλό. Από την άλλη όμως έχουμε το ζήτημα της ιδιοκτησία των δεδομένων. Σε ποιον ανήκουν. Οι αστρονόμοι για παράδειγμα συλλέγουν πάρα πολλά στοιχεία και τα βγάζουν στο διαδίκτυο. Τα δημοσιεύουν και τα χρησιμοποιούν διάφοροι άλλοι για να τα αναλύουν. Ε, και ε, προχωρούν σε νέες ε, ε, γνώσεις, σε νέες ανακαλύψεις, τις οποίες και δημοσιεύουν. Δηλαδή τα στοιχεία συλλέγονται και αναλύονται. Εάν εμείς αυτό το αποτρέψουμε δεν υπάρχει πρόοδος. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι η αυτοματοποίηση. Θα ήθελα να παρακαλέσω τα μέλη του πάνελ να ε, έρθουν στα εργοστάσια να δούνε πώς παράγονται αυτόματα κάποια υλικά όπως είναι το γυαλί. Ε, βλέπουμε από τη μια λοιπόν τις μετρήσεις, ε, τη συλλογή των στοιχείων στην αλλουργία. Ξέρετε πώς γίνεται το γυαλί με άμμο και διάφορες άλλες πρωτεσίλες. Και από την άλλη ε, είναι αυτόματη η διαδικασία παραγωγής. Όλα ρυθμίζονται, όλα έχουν πρωτόκολλο, παντού συλλέγονται δεδομένα και αποθηκεύονται σε συγκεκριμένα σημεία. Υφίστανται λοιπόν μια επεξεργασία και μετά ανάλογα με τις απαιτήσει έχουμε ε, διάφορα μεγέθη γυαλιού που κόβονται και ε, συναρμολογούνται. Και εδώ μιλάμε για βιομηχανία 4.0. Το ίδιο ισχύει και για ε, το γυαλί που χρησιμοποιείται ως ε, συσκευασία. Οι άνθρωποι εκεί είναι μηχανικοί, είναι προγραμματιστές, είναι ε, ειδικοί ε, ε, πληροφορικής που αυτά τα εφαρμόζουν από την αρχή στη μέση και το τέλος της παραγωγής. Αυτή είναι η κανονική διαδικασία παραγωγής ε, σε ένα εργοστάσιο. Και στο Ινστιτούτο Φρανχόφερ μπορείτε εσείς να εργάζεστε για να προετοιμάζετε το μέλλον, αλλά δεν έχετε και πάρα πολλά καινούρια να εφεύρετε σε σχέση με αυτό. Ερωτώ λοιπόν, θεωρείτε ότι είναι σωστό να έχουμε ένα ενιαίο πρωτόκολλο για τη συλλογή των δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ντάριο Ταμπουράνο από το ε, <clears throat> Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους γιατί μας αναπτύξατε διάφορα σενάρια για το πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στο μέλλον. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία των νέων τεχνολογιών. Σε σχέση με τον ομιλητή της Siemens, θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα. Θα ψηφίσουμε αύριο μία έκθεση για την ενεργειακή σήμανση. Τι πιστεύετε λοιπόν για τις ευφύς συσκευές. Εδώ μιλάμε για τις ε, οικιακές συσκευές γενικότερα και τι πιστεύετε για την χρήση των smartphones. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποια είναι τα στοιχεία χρήσης και κατανάλωσης, έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να είναι αποδοτικά για μία ποιοτική αποτίμηση και να μειώσουμε το κόστος χρήσης για τον ε, τελικό χρήστη. Πώς έχει κατάσταση σε άλλες υπήρους όπως την Ασία και την Αμερική. Ε, πώς βλέπουν το θέμα οι νομοθέτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Επόμενος. Ο μιλητής ήταν ο κύριος Ρόιλ, ο οποίος αποχώρησε, αλλά ο Εδουάρ Μαχτά έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Ακούγοντας όλες τις παρεμβάσεις, είναι σαν ε, να, γίνονται τα έργα επιστημονικής φαντασίας πραγματικότητα. Ένας επιχειρηματίας που κάθεται σε ένα γυάλινο ουρανοξύστη στην Νέα και πατάει ένα κουμπί και γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Ποιο όμω θα πληρώσει το κοινωνικό μοντέλο είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το απαντήσουμε γιατί και αυτό θα έχει έναν αντίκτυπο. Αυτή η βιομηχανία 4.0 ε, σίγουρα αυξάνει και τον εξεχωρισμό. Ε, μας είπατε διάφορα και όλα αυτά θα μας βοηθήσουν και στις συζητήσεις που έχουμε αυτό τον καιρό. Γιατί κανείς δεν θα μπορέσει πλέον να μας ε, πείσει ότι είναι δύσκολο, πολύπλοκο ή αδύνατο να έχουμε την ιχνηλασιμότητα ε, προϊόντων που παράγονται όπου και αν παράγονται. Γιατί έχουμε τώρα μια συζήτηση για το ETS και όταν ε, εγώ ζητώ κάποια πράγματα πλέον ένα προϊόν που έρχεται από την Κίνα πώς θα το εντοπίζουμε, τι, τι πόρη έχει ακολουθήσει. Να εσείς μας απαντάτε και την είναι αυτά. Αυτή η βιομηχανία 4.0 θα είναι χωρίς ανθρώπους, άρα για ποιον. Και τέλος, η επιτάχυνση καλή είναι, αλλά τα δίκτυα, το είπαν και κάποιοι, είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες αυτού του βιομηχανία 4.0. Ε, Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε για τα σχόλιά σας αλλά και τις ερωτήσεις σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε κανέναν άλλο εκτός από τον κύριο Μπόνη. Αν δεν θέλει κανείς άλλος θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπόνη. αν δεν θέλω λέει ο κύριος Μπόνη. Μα ήρθε η ώρα σας. Αφού σας διέκοψα προηγουμένως και θέλετε να τελειώσετε. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε, με κάλυψαν οι συνάδελφοι. Ήθελα να ρωτήσω τι είδου κανονισμού χρειαζόμαστε, ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο και το μη κανονιστικό πλαίσιο που χρειάζεται για τι λύσει αυτέ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και έχει σημασία να κατανοήσουμε. Σε πολλούς τομείς, λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ τη νομοθεσία και τη τεχνολογία. Ε, πάντα μοιραία θα ε, κερδίζει η τεχνολογία, γιατί τρέχει με πιο ραγδαίους ρυθμούς από ότι ο κόσμος μας και η νομοθεσία μας. Οπότε έχει νόημα να το καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε σε κάποιους τομείς κανόνες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ισχυρή νομοθεσία πάντα. Και θα πρέπει να δούμε σε ποιους τομεί ε, θα χρειαστεί νομοθεσία και πού όχι. Υπάρχει η λεγόμενη ήπια νομοθεσία. Ε, οι εθελούσει ρυθμίσεις, η αυτορύθμιση, οι κώδικε διοντολογίε, νομίζω τα λένε κάπως έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Όταν όμως συζητούμε για κάποια κρίσιμα ζητήματα και κλειδιά λύσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κείμενη νομοθεσία. Ε, σε σχέση με αυτό το θέμα της ευθύνης των ρομπότ δεν είναι απλέ οι λύσεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έμπνευση που είχατε να μας τα παρουσιάσετε όλα αυτά και ε, την, ε, την έννοια ε, του ηλεκτρονικού προσώπου. Κατανοώ ότι και εσείς τηρείτε τις αποστάσεις από την έννοια αυτή και είναι πολλά τα ερωτηματικά. Αλλά βήμα-βήμα θα πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι το πλαίσιο που χρειάζεται, το κανονιστικό και πώς θα υποστηρίξουμε τις εξελίξεις. Το ανέφεραν και οι συνάδελφοι προηγουμένω και με κάλυψαν, οπότε αυτή η μικρή προσθήκη μου. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να ε, επανέλθουμε τώρα στους ομιλητές μας για να απαντήσουν. Δεν ξέρω αν θέλετε, έχουμε χρόνο να απαντήσετε, παρακαλώ. Πρώτος ο κύριος Ρούλαντς. So I... Πολλές ήταν οι ερωτήσεις, τις ε, κατέγραψα, αλλά δεν ξέρω αν τις έχω ε, καταγράψει όλες. ως προς τον κύριο Μαρτέν, δεν νομίζουμε ότι θα απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τα εργοστάσια. Στο Αμβούργο είχαμε ε, ένα εργοστάσιο όπου συμμετείχαν 1.200 εργαζόμενοι και τώρα είναι μία ε, βιομηχανία τύπου 4.0, αλλά υπάρχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, ο ίδιος αριθμός. Δηλαδή, τι γίνεται, καταρτίζονται και εκπαιδεύονται ανάλογα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Εάν δεν το είχαμε κάνει αυτό, τότε το εργοστάσιο θα είχε κλείσει σήμερα, γιατί δεν θα ήταν ανταγωνιστικό. Άρα το θέμα είναι να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί με τον υπόλοιπο κόσμο και πρέπει κανείς να ακολουθήσει τις τάσεις που διαγράφονται. Αλλιώ θα το κάνουν στην Κίνα, στην Νότιο Κορέα και αλλού. Αν δείτε τη ε, ρομποτική έχει διενεργηθεί μία μελέτη όπου η, Γερμανία έχει βγάλει. 380 ρομπότ ανά 10.000 ενώ η Κορέα έχει 300, η Ιαπωνία 400 και ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 80 ρομπότ. Αν γίνεται λοιπόν στην Ιαπωνία, Κορέα και ΙΠΑ θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την τάση. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν είδαμε μείωση του εργατικού δυναμικού στο Αμβούργο, σε αυτό το πλέον σύγχρονο εργοστάσιο. Σε σχέση με τη χρήση των δεδομένων και βελτιστοποίησή τους, στο τέλος έχουμε το ίδιο μοντέλο όταν χρησιμοποιήσουμε αυτή την αλυσίδα παραγωγής ε, για τα, τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων, χρησιμοποιούμε τους ίδιους αλγορίθμους, αλλά θεωρούμε ότι οι καταναλωτές βλέπουν ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς, ε, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα BMW, Porsche, Maserati. Παρόλα αυτά υπάρχει μια ειδική τάση και στο σχεδιασμό και στην όλη αλυσίδα παραγωγής. Άρα αφήνουμε την αγορά να δράσει. Ως προς τα πρότυπα τυποποίησης και τον περιορισμό τους, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει παγκόσμια τυποποίηση και να συνδυαστεί με μια ήπια νομοθεσία, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να προσαρμοζόμαστε άμεσα, τάχιστα στις αλλαγές. Διαφορετικά θα βρεθούμε εκτός νυμφώνους. Σε σχέση με τη συνδεσιμότητα, ναι, πράγματι χρειάζεται υποδομή και για τη βιομηχανία 4.0 χρειάζονται και ευρυζωνικά συστήματα, η χρήση τους δηλαδή. Δηλαδή έχει σημασία και η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. Θα πρέπει να είναι υψηλότερη δυνατή, κάτι το οποίο δεν ισχύει παντού στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, υψηλής ποιότητας δίκτυα. Θα παραμείνω εδώ για να πάρουν το λόγο και οι άλλοι συνάδελφοι. Ναι, και μπορείτε να προσθέσετε κάτι στο τέλος. Προς τον κύριο Κάκελάινεν υπήρξαν ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σε σχέση με τη συνδεσιμότητα, ε, εδώ αυτός ο τομέας μας απασχολεί, χρησιμοποιούμε αυτούς τους ε, αισθητήρε και έχουμε έχουμε και μία παγκόσμια συμφωνία περιαγωγής με ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο δίκτυο. Έχουμε τις ίδιες ε, ε, εμπορικές δραστηριότητες με αυτές που υπάρχουν στον τομέα της κινητής ε, τηλεφωνίας, όπου υπάρχει η συνδεσιμότητα δεδομένων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από τα έξοδα περιαγωγής και να φτάσουμε σε μια κοινή τεχνολογία, μια κοινή πλατφόρμα για την συνδεσιμότητα που θα λειτουργήσει σαν πλατφόρμα για την καινοτομία, την τεχνολογία, έτσι ώστε και οι μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες και να συλλέγουν περισσότερα δεδομένα σε μάλλον δέκα χρόνια πριν, όλοι οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών ήθελαν να ανελιχθούν στην ε, αλυσίδα αξιών για να έχουν ε, περισσότερες πωλήσει. Τώρα, ε, ως προς τα δίκτυα αυτά, βλέπουμε ότι οι φορείς τηλεπικοινωνιών προσπαθούν να χτίσουν τα δικά τους ε, δίκτυα για να μπουν σε αυτή την αλυσίδα αξιών. Έτσι ώστε η δικτυακή συνδεσιμότητα να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ε, αυτή τη νέα τεχνολογία των ε, πολλαπλών αισθητήρων. Επίσης μιλήσαμε για το δημόσιο έναντι του ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ότι τα στοιχεία που συλλέγονται από δημόσιους φορείς θα πρέπει να είναι δημόσια. Και ιδιαίτερα τα πρώτα στοιχεία, τα πρωτογενή στοιχεία τα οποία συλλέγονται. Θα πρέπει όμως να τα επεξεργαστούμε για να φτάσουμε στη σωστή πληροφορία. Χρειάζονται αναλύσεις, αλγόριθμοι και ούτω καθεξής. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι μια δημόσια διεργασία, ανοιχτή δηλαδή παρουσίαση, γιατί μιλάμε για παροχή υπηρεσιών και τεχνολογίας. Αυτό μας ενδιαφέρει στην κοινωνία, δηλαδή να υπάρχουν επιχειρήσεις και να δίνουν δουλειά στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Ε, ευχαριστώ ε, κύριε Κακελάινεν που είστε διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΕΟ. Ε, θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ματίας Πούτσα από το Ινστιτούτο Φράουνποφερ. Κυρίε και κύριοι, καταρχά δεν θα σα ζητήσω συγγνώμη που είμαι καθηγητή στο Φρανκόφερ και κάνω έρευνα. Δεν θα ζητήσω και συγγνώμη και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν είμαι πολιτικό. Γιατί να σα πω το εξή ό,τι και να κάνετε με τη βιομηχανία 4.0, κάντε το γρήγορα, διπλάσιο και τριπλάσιο χρόνο από ό,τι προτείνουμε. Γιατί ε, ε, ζούμε σε έναν κόσμο που το θέμα αυτό δεν είναι απλώ θέμα συζήτηση φιλολογική, Και θυμάμαι πριν από πέντε χρόνια ε, το Φράουνχόφερ μίλησε ε, ε, για τα τρία γιώτα στα αγγλικά, ε, για τη συμμετοχή που θα είναι ο κόσμος με τη γενοτομία κτλ. Και το τρίτο γιώτα ήταν involving people, να συμμετέχει και ο κόσμος. Γιατί όλοι εδώ οι νέοι που κάθονται στα πίσω έδρα να εργάζονται εδώ. Εγώ είμαι περίπου 55 και κάτι, εν πάση περιπτώσει. Και έμαθα να χρησιμοποιήσω ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο οι νέοι μας χρησιμοποιούν αυτόματα, γιατί αυτό το γνωρίζουν. Ε, και αυτά θα έρθουν λοιπόν, η τεχνολογία μας ξεπερνάει. Και οι μεγάλες εταιρείες και οι Siemens τώρα δημιουργούν, λέει, καινοτομία και hubs για νεοφυείς επιχειρήσεις, γιατί γνωρίζουν ότι η καινοτομία ε, σε ένα μεγάλο οργανωμένο σύστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Και πέρα λοιπόν από τις μεγάλες εταιρείες δημιουργούν συστήματα καινοτομίας. Πρώτα λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, κάντε το γρήγορα και κάντε το ε, για χρήση. Γιατί συνήθως ε, αυτοί που παίρνουν αποφάσεις είναι 45 ετών και πάνω και έμαθαν το κινητό να το δουλεύουν από τα παιδιά τους και όταν χαλάσει το δίνουν στο γιο τους ή στην κόρη να το φτιάξει. Απαντώ τώρα στην κυρία Βέρνερ στα αγγλικά. Ε, έχετε και όταν δημιουργήσαμε αυτό ε, το κέντρο έρευνας πριν από τρία χρόνια η πρώτη ε, επίσκεψη ήταν από συνδικάτο που μας θύψε την πόρτα και μας λέει για ελάτε εδώ εσείς τι κάνετε. Ε, τώρα έχουμε την ευκαιρία, πριν από 25 χρόνια, όταν αρχίσαμε ε, στην ε, τεχνολογία των κατεργασιών μας, λέγανε δεν έχετε τα συστήματα, ο επιταχυντής είναι πολύ γρήγορος, είναι πολύ περίπλοκος, δεν έχουμε τα δεδομένα και βάση περιπτώσει. Έγινε τώρα και έχουμε 100% προσωμείωση διαφόρων κατεργασιών. Το ίδιο θα ισχύσει και με τα δεδομένα και θα ισχύσει. Και το ενδιαφέρον είναι να βρεις ανθρώπους που ε, έχουν συνηθίσει να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά και είναι θέμα ευελιξίας αυτό. Και κύριε Κόχλιτσεκ, αυτό που μας εξηγήσατε για την ε, η είναι 100% αυτοματοποίηση, δεν είναι 4-0, δεν είναι το νέο επιχειρηματικό μοντέλο, επιχειρησιακό μοντέλο. Το θέμα είναι να εξηγήσετε στον κόσμο ότι όταν έχει πέντε χρόνια χρησιμοποιήσει το γυαλί, τι να το κάνει μετά για να το ανακυκλώσει. Αυτό που κάνετε εσείς είναι αυτοματοποίηση. Και κύριε Μπιουτικόφερ για την Κίνα, εκπλήσουμε λίγο. Σκέφτηκε ποτέ κανείς ότι αυτό δεν θα συνέβαινε με την κουπκά, με τα ρομπότ, τα κινέζικα. Στο δικό μας πανεπιστήμιο, στο Χέμνιτς, στο Πολυτεχνείο, έχουμε 10% ξένους φοιτητές, οι περισσότεροι είναι Κινέζοι. Και σήμερα είναι λίγο πολύ τα παιδιά ε, των πλουσίων. Δεν είναι και τα πιο λαμπρά μυαλά. Φανταστείτε να έρθουν τα πιο λαμπρά κινέζικα μυαλά στο Χέμνιτς. Αλλά αυτό είναι η βασική η κανονική διαδικασία. Θα πρέπει να το μάθουμε και να γίνουμε εμείς πιο γρήγοροι και πιο καινοτόμοι. Και ήταν και δική μου ιδέα αυτό, ε, με αυτό τον κύκλο που σας έδειξα. Ε, δεν ήσασταν εδώ όταν τα έλεγα κύριε Μπιουτικόφερ. Δεν είναι νόμος της φυσικής ε, δεν έχουμε εφευρέσεις να πούμε ότι ε, τα κομπιούτερ μας δεν είναι αρκετά γρήγορα. Όλα αυτά συμβαίνουν. Ναι. Δεν καλούμαστε να ανακαλύψουμε τίποτα. Απλώς θα πρέπει να γεμίσουμε το κενό με τις ε, δυνάμεις μας, με τα καινοτόμα σχέδια, με τις νέες ιδέες και τα δίκτυα. Θα συμβούν όλα αυτά. Για δύο λόγους έχουμε να μάθουμε ε, ε, από την Κίνα, να μάθουμε από αυτούς και να πάμε ως γερμανική βιομηχανία και ευρωπαϊκή στην Κίνα. Αυτά τα δύο κάνουμε. Στρατηγική, κανονική δεν έχουμε για την Κίνα. Θα τα βρούμε μπροστά μας όμως όλα αυτά. No, Αυτός ήταν ένας τρόπος με πάρα πολλές λέξεις για να μας πείτε ότι όχι στρατηγική δεν έχουμε. Ακριβώς. Ε, ωραία. Παρακαλώ, απαντήσει ε, τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Πέτερ Μπρόιτιγκα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να σας ενθαρρύνω γιατί εσείς είσαστε εδώ ε, στο σωστό μέρος. Δεν είναι πλέον εθνικό το ζήτημα. Είναι διεθνές. Τουλάχιστον ευρωπαϊκό. Σκεφτείτε τις συζητήσεις ε, για την ε, ασπίδα τη θωράκιση προσωπικών δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Ένωση, το Privacy Shield. Χρειαζόμαστε ισχυρή ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε για το τι είδου νομοθεσία μιλάμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, μην ε, καταλήξουμε σε υπερρύθμιση και συμφωνώ με του προλαλήσαντε. Ναι, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως πολύ προσεκτικά να δούμε πού και τι θα ρυθμίσουμε. Ας έλθω στην κυριότητα των δεδομένων πρώτα απ' όλα. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, γιατί εδώ δεν έχουμε ένα κόνσεπτ. Δεν είναι όπως ο νόμος περί δικαιωμάτων δημιουργού, πνευματικών δικαιωμάτων, αθέμητων εμπορικών πρακτικών και ούτω καθεξής. Είναι ένα κομματάκι, ένα μικρό μέρος της πίτας αν θέλετε και γιατί πρέπει να το προστατεύσουμε μπορεί να παράγεται τυχαία από μηχάνημα από αυτόν που έχει λεφτά για να χειρίζεται ένα μηχάνημα και ούτω καθεξής γιατί πρέπει να το προστατεύσουμε για ποιο λόγο πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά κατά πόσον χρειαζόμαστε ε, κυριότητα δεδομένων θα μπορούσαμε ίσως να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να έχουμε ένα κανονισμό για την πρόσβαση στα δεδομένα γιατί έχουμε δεξαμενές δεδομένων και ίσως θα ήταν καλό να ρυθμίζεται η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα με κάποιο κανονισμό. Αλλά και αυτό είναι δύσκολο, διότι υπάρχει δέσμη ευρωπαϊκών κανόνων για το θέμα αυτό, εμπορικό απόρριτο, βάση δεδομένων, ιδιωτικότητα δεδομένων. Υπάρχουν κανονισμοί λοιπόν που είναι μια χαρά και ίσως θα μπορούσαμε αντί να έχουμε τη μεγάλη έκρηξη, ένα big bang για ε, μια νομοθεσία σε σχέση με τα μαζικά δεδομένα, να εστιάσουμε στις οδηγίες που έχουμε ήδη, στις διατάξεις που ήδη ισχύουν, για να μην υπερρυθμίζουμε τα πράγματα και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Συμφωνώ επίσης με τον Φιλανδό, ομιλητή που είπε ότι οι κυβερνήσεις σας πληρώνουμε τόσους φόρους. Ίσως θα μπορούσαν τα δεδομένα να είναι ανοιχτά, open data, να τα έχουν όλοι κτλ. Για τι επιχειρήσει όμως που έχουν εργαστεί σκληρά για να αποκτήσουν πλεονέκτημα, αν τους πει κανεί, πρέπει να ανοίξετε όλα τα δεδομένα πέραν το εμπορικό, κτλ., τα είναι ίσω λίγο υπερβολικό. Google, Facebook δεν το κάνουν. Δεν είναι open data για όλου τα δεδομένα αυτών των δύο στο σύλλογο. Ας μην υπερβάλλουμε. Δεύτερον, ευθύνη. Έχει να κάνει με το εθνικό δίκαιο. Με την ψηφιοποίηση όμως δεν θα ισχύει αυτό πια. Γι' αυτό και εσείς είπα, είστε στη σωστή θέση εδώ για να μιλήσετε για την ψηφιακή ευθύνη, όχι μόνο την ευθύνη των ψηφιακών αγαθών, αλλά για την ψηφιοποίηση και το βιομηχανία 4.0. Δεν μιλάμε πια για τη Γερμανία, τη Ρωσία, την Ελλάδα. Δεν είναι πρόβλημα εθνικό, είναι ευρωπαϊκό. Επομένως, πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε ίσως νέες έννοιες και αυτό μπορεί να σημάνει την αρχή για ένα ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο ενδεχομένω, ξεκινώντα από την ψηφιοποίηση. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί και προσωπικά δεν πιστεύω ε, ότι μπορούμε να έχουμε μία λύση εύκολη με, νέο, ε, με κάποιο νέο κόνσεπτ. Για δείτε στη Γερμανία ένα σύστημα μπορεί να δουλεύει 120 χρόνια. Γιατί να το καταλήψουμε με τη μία. Γιατί να μην δούμε τι συστήματα υπάρχουν στην Ευρώπη, στη Γαλλία και αλλού και από εκεί πέρα προχωρήσουμε. Επομένως, εγώ δεν είμαι υπέρ του να έχουμε άμεσα το ηλεκτρονικό πρόσωπο. Σε κάποιο μεταβατικό στάδιο, ναι, όχι άμεσα όμως, γιατί αν πρέπει άμεσα να το ρυθμίσουμε θα πρέπει να σκεφτούμε τόσα πολλά πράγματα και δεν τα γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Για τις εφευρέσεις υπάρχει αρχή. Ας περάσουμε το ρουβίκονα όταν έρθει η ώρα του. Αλλά μην ε, ε, το παρακάνουμε τις θεωρητικές συζητήσεις. Αλλά τέλος πάντων, ε, εγώ είμαι εδώ ως δικηγόρος. Το επόμενο σημείο στρατηγική. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι δεν έχουμε στρατηγική και είναι κρίμα. Γιατί αν χρηματοδοτούνται επιστημονικά έργα, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με κονδύλια από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με κονδύλια των φορολογουμένων, νομίζω ότι θα πρέπει οι εφευρέσεις με διανόμου να ορίζεται ότι θα παραμένουν στην Ευρώπη και όχι ε, να παραχωρούνται στην Κίνα ή αλλού. Ε, τώρα έβγαλα το καπέλο του δικηγόρου και έβγαλα το καπέλο του πολιτικού. Και τέλο, ναι, για το εργασιακό δίκαιο, πολύ σημαντικό ζήτημα. Έχει γίνει έρευνα. Τεράστιο το καθήκον μα για την μεταφορά του εργατικού δυναμικού θα υπάρχει δουλειά, αλλά θα είναι διαφορετική. Και αυτή η μεταφορά, η μετατόπιση είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Και αυτό τον καιρό συζητείται και κάτι ακόμη. Όλα αυτά πώς θα χρηματοδοτηθούν και αν υπάρχει λόγος να χρηματοδοτηθούν. Και επειδή τα ρομπότ κάνουν τη δουλειά, τελικά χρηματοδοτούνται όλοι από το κράτο. Το έχουμε συστήσει και αυτό. Δεν είναι αυτό ο σωστός τρόπο. Πρέπει να υπάρχει εργασία, αλλά να είναι αμοιβόμενη αυτή η εργασία. Και να είναι πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα μετάβαση. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και η νομική επιστήμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους σας. Πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλια, οι ομιλίες. Και ε, Σας ευχαριστούμε που μας ήρθατε και να μας ξανάρθετε του χρόνου, δεν ξέρω πότε. Αν θα έχουμε τελειώσει όλη την νομοθεσία, αν είμαστε αρκετά γρήγοροι και πάλι σας ευχαριστώ. now, uh, we will start Και τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 10 λεπτών ίσως για να προχωρήσουμε στην Επόμενη έκθεση που είναι του συναδέλφου Φέντερλε. Αλλά να ακούσουμε πρώτα τι έγινε στο Κόρκ. Να μας πει ο κύριος Ζανονάτο για την αποστολή στην Ιρλανδία. Άρα όχι διάλειμμα. Πράγματι ήταν μία άκρος ενδιαφέρουσα αποστολή αυτή της Ιρλανδίας το Μάρτιο. Συμμετείχαμε τους Ρούμπιχ, Κέλ, Πούσεκ και Κάπελ. Θα ήθελα να πω ότι όλες οι συναντήσεις ήταν άκρος ενδιαφέρουσες. Είδαμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που βρίσκεται στην εμπροστοφυλακή της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί απασχολούμενοι σε αυτό τον ε, τομέα. Στο Tindal National ε, Institute στο Κόρκ έγινε η πρώτη συνάντηση. Ο Τίνταλ ήταν, ε, ένα, ήταν ένας μεγάλος επιστήμονας και είναι ο πρώτος που ανακάλυψε τα αέρια θερμοκηπίου. Ε, μιλήσαμε λοιπόν για θέματα που άπτονται της ε, επικοινωνίας και ο Ρόναν Μαρφή μίλησε για άμεση συνδεσιμότητα μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Ο ακαδημαϊκός κόσμος της Ιρλανδίας συνεργάζεται στενά με τις επιχειρήσεις και αυτό και για το υπολογιστικό νέφος και την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Ο καθηγητής Σάλιβαν μας μίλησε για την ανάγκη δημιουργία μιας μάγνα κάρτα για τα δεδομένα και για την προστασία των δεδομένων έτσι ώστε να ε, γίνουν κοινωνοί των εξελίξεων και οι επιχειρήσεις αλλά και η κοινωνία των πολιτών μετά επισκεφτήκαμε το Cork Institute of Technology, όπου είδα ότι χρησιμοποίησε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και τον ορίζοντα 2020 για τα ενεργειακά προγράμματα και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, επισκεφτήκαμε Είκαμε το Θαλάσσιο Κέντρο Έρευνας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ιρλανδία μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενέργεια που ε, μπορεί να δημιουργηθεί με βάση τα παλιροϊκά κύματα και έχει πραγματικά εκμεταλλευτεί αυτό το τομέα. Επίσης στο Σάνον επισκεφτήκαμε τον σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου και παρά το γεγονός ότι αυτό το σχέδιο είναι κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, είναι πολύ δύσκολο για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να περιλαμβάνουμε προγράμματα ύψης της σημασίας, κάτι όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη ε, εξέλιξη του τομέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για τη διοργάνωση αυτής της αποστολής. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Θα ήθελε κάποιος να ρωτήσει, κάτι να προσθέσει. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και να σας συγχαρούμε για αυτή την ε, άκρος ενδιαφέρουσα εργασία και τις επισκέψεις. Και τώρα προχωράμε με την επίσκεψη στη Φιλανδία και στην Εστονία. θα ήθελα ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Φιλανδίας να μας ε, μιλήσει για την εξέλιξη. Καταρχήν σας ευχαριστώ. Για... Ευχαριστώ πολύ για, καταρχάς για τη συμμετοχή σε αυτή την επίσκεψη. Όσους ήρθαν να ευχαριστήσω τον Μάρκε και τη Γραμματεία κυρίως ήταν πάρα πολύ καλή η επίσκεψή μας. Πήγαμε πρώτον στο Φινλανδικό Κοινοβούλιο, είπαμε ότι αποφάσεις λαμβάνονται ε, με πολύ δημοκρατικό τρόπο. Υπάρχει Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ε, στην οποία λογοδοτούν και οι Υπουργοί. Είναι κάπως διαφορετική η διαδικασία σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης ε, έχουμε το FES δίκτυο και το Εθνικό Δίκτυο, FinGrid, Πήγαμε λοιπόν εκεί και μιλήσαμε για ένα πρόγραμμα για την ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά την αγορά λιανικής πόλης ηλεκτρικού ρεύματος. Και όλοι οι φορείς έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Εύκολα μπορεί κανείς να αλλάξει προμηθευτή ή διεύθυνση. Προμηθευτές καταναλωτές λοιπόν όπως είπα Ησυχία, δεν ακούω τη φωνή μου παρακαλώ. Is, is with the start. Νεοφύς ναι, επιχειρήσεις ήταν το τρίτο. Πήγαμε στη σάουνα και μια άλλη επιχείρηση τεχνίων. Η σάουνα, για παράδειγμα, έχει εργαστεί με 160 επιχειρήσεις από τη Σκανδιναβία, από τη Ρωσία και από την Ανατολική Ευρώπη και έχει προγράμματα σε διάφορες χώρες. Και είδαμε και την ΤΕΚΕΣ ε, για την έρευνα και ανάπτυξη που χρηματοδοτεί πολλές δραστηριότητες, ιδίως νοφίες νεοφυείς επιχειρήσεις. Τώρα, αυτό ήταν την τρίτη, την πρώτη μέρα. Στη δεύτερη μέρα, την τετάρτη, είχαμε μια κοινή επίσκεψη Ένβη και Ήτρε. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλο προηγούμενο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο που ήταν η Ένβη και μαζί. Πήγαμε στο δάσος, και μιλήσαμε για την βιοοικονομία. Δεν χωριστήκαμε να μιλήσουμε δηλαδή από τη μια για την κατομία από την άλλη για το περιβάλλον, αλλά τα είδαμε από κοινό αυτά τα θέματα. Πήγαμε λοιπόν εκεί και είχε έρθει και ο κλάδος της νοσοκομείας. Ελπίζω να θυμάστε όλοι ότι δεν έχει μείνει ε, αναξιοποιητό κανένα ε, τμήμα του δάσους. Μέχρι κίνες έχουμε τις επελέτες, έχουμε τα ροκανίδια, όλα χρησιμοποιούνται. Όλα τα πρώτα της υλοτομίας χρησιμοποιούνται. Είδαμε και τα περιπιστοποίηση των προϊόντων δασοκομείας και μετά είδαμε την Ομοσπονδία Χημικής Γεωμηχανίας ε, και την Πετρελαιομηχανία. 2,5 εκατομμύρια μόνο τόνοι είναι ανανεώσιμες πηγές, πολύ περισσότερο το πετρέλαιο. Θέλουμε να εστιάσουμε όμως στην χλασιμότητα, στη βιωσιμότητα. στις ανανεώσιμες ε, όταν έχουμε ε, φυτικά έλαια υπάρχει η χνηλασιμότητα. Δεν είναι το ίδιο όμως με τη βιομηχανία τροφίμων. Στην έρευνα και ανάπτυξη απασχολούνται χιλιά άτομα. 70% των εταιριών εστιάζουν στις ΑΠΕ. η Λουφθάνσα και τα λοφόρια του Σαν Φρανσίσκο χρησιμοποιούν τα καύσιμα αυτά μάθαμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Έπειτα πήγαμε στο Ταλίν με το πλοίο. Είδαμε πολλά. Υπάρχει ένα νέο εργοστάσιο για μάλλον ένα, ένα πηγείο που θα φτιάχνει ένα πλοίο που θα μπορεί να ε, φιλοξενεί 40% περισσότερους επιβάτες θα επιταξιδεύουν από, την, από το στο Ταλίν και θα εξοικονομεί ενέργεια. Στη Βάρτσιλα Μότορς τώρα κάναμε επίσης μια επίσκεψη. Είναι παραγωγή κινητήρων ε, για την αυσπλοεία, κυρίως ε, ε, ειδικεύονται στους κινητήρες που χρησιμοποιούν ε, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Μιλήσαμε επίσης για το διοξίδιο του θείου, για τα ζωτούχα και άλλα ε, αέρια. Με το LNG θα πέσει πολύ και η, η ρήπανση. 90.000 είναι ο τοπικός τόλος. 119 μόνο τα ε, κινούμενα με φυσικό αέριο και πολύ μεγάλο ποσοστό παράγεται από τη Βάρτσιλα Μότος. Μάθαμε πολλά για την απήγηση, για την προμήθεια LNG. Η Ήτρε νομίζω ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα όλα τα μέλη. Έπειτα Είχαμε και την εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαίσιου που θέλαμε να συζητήσουμε. Μετά στην Εστονία πάντα την επόμενη μέρα πήγαμε στο Κοινοβούλιο, είδαμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων που ουσιαστικά ακολουθούν την ίδια διαδικασία με, την, με το Φινλανδικό Κοινοβούλιο και μιλήσαμε και με τους οδηγούς ταξί Uber. Εκεί ρυθμίζεται το θέμα, στην Εστονία συγκεκριμένα. Είναι η πρώτη ανάγνωση, τώρα ετοιμάζει τη δεύτερη ανάγνωση. Από την πρώτη φορά που χρησιμοποιήσει κάποιος ε, την υπηρεσία Uber πληρώνει και κοινωνική ασφάλιση για τους οδηγούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγαμε και στο Estonia Showroom ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ε, ευρωπαϊκή θαγένεια. Δύο εκατομμύρια στον Ή θέλουν ε, δέκα εκατομμύρια ηλεκτρονικούς πολίτες όμως. Όλοι οι Εστονοί έχουν επίσης ένα δημόσιο λογαριασμό και με αυτήν την ταυτότητα έχουν υπηρεσίες από πάρα πολλές ε, εταιρείε δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης συζητήσαμε κάποια θέματα που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία και την ενέργεια. Αυτά και ευχαριστώ όλους ε, που ήταν στην αποστολή αυτή. Μπορείτε να διαβάσετε και πιο αναλυτικά το έγγραφο. Ευχαριστώ πολύ. Λέω πρόεδρος, υπάρχουν σχόλια. Υπάρχει κάτι που θα θέλετε να προσθέσετε. Όχι, κανείς δεν θέλει να πει τίποτα. Σας ευχαριστώ για όσα κάνετε λοιπόν και στη δική σας χώρα τη Φιλανδία αλλά και στην Εστονία. Επόμενος με τις μέρες διάταξης. Οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών και το αποτυπώματος άνθρακα. Πολύ σημαντικό θέμα. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Συντάκτης γνωμοδότησης ο Φρέντρικ Φέντρλε. Δυνάμει του κανόνος 54. Ενισχυμένη συνεργασία. Συντάσσεται αυτή η γνωμοδότηση. Παρίστατες λοιπόν ο συντάκτης μας σε όλες τις συνεδριάσεις των σκιωδών της ΕΝΒΗ και στους τριλόγους θα συμμετάσχει. Βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει μας περισσότερο είναι η διαρροή άνθρακα αφενό και τα κονδύλια, τα ταμεία αφετέρου. Αλλά βέβαια οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να το αναφέρετε σε αυτή τη συζήτηση. Απλά αυτή είναι η δική μας αρμοδιότητα. Ας το συζητήσουμε όμως. Να ζητήσω από τον εισηγητή πρώτα απ' όλα να λάβει το λόγο. Φρέντρικ, σε ακούμε. Ευχαριστώ. Καταρχήν, χαίρομαι που γίνεται έγκαιρα αυτή η συζήτηση. Είναι τεράστιο το θέμα και έχει μεγάλη σημασία να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση με τις πολιτικές ομάδες για να δούμε αν υπάρχει διαφάνεια και να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση. Έχουμε μέχρι Τετάρτη την προθεσμία για υποβολή τροπολογιών στην έκθεση μου. Ε, υπάρχουν ορισμένε κατευθυντήριες γραμμές που ακολούθησα ασχολήθηκα με το όλο θέμα μέσα στα πλαίσια της ε, αρμοδιότητας, της κύριας αρμοδιότητας της Επιτροπής ε, Ήτρε. Και πάντα έλεγα προς τους σκιώδεις ότι υπάρχουν ε, ορισμένες αρχές πέρα από ζητήματα τεχνικού χαρακτήρα. Α, όταν το Σεπτέμβριο όμως ε, φτάσουμε σε μια πλειοψηφία, το ελπίζω τουλάχιστον, θα γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Ε, καταρχήν δεν πρέπει να προωθήσουμε το ε, συντελεστή διόρθωσης, γιατί από όσο ξέρω θα χάσουμε ένα 17% ε, ε, αυτό θα είναι το επιτρεπτό όριο, δηλαδή με βάση το 100 θα χάσουμε 17, δηλαδή θα φτάσουμε το, στο 83%. Είναι και η μακρύτερη περίοδος για την ανταλλαγή εκπομπών. Άκουσα ορισμένους συναδέλφους να λένε ότι υπάρχει ένα ε, ίσο δικαίωμα να έχουμε, υπάρχουν ίσα δικαιώματα ως προς τα επιτρεπτά όρια. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε να φτάσουμε σε κάτι σαν την ΚΑΠ για τον βιομηχανικό τομέα με βάση την ελεύθερη αγορά. Η το σχέδιο διαρροής του άνθρακα θα έπρεπε να λήξει σε, αυτό, σε αυτή τη φυτεία, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα όρια στην αγορά είναι περιορισμένα και δεν θα πρέπει να πιέσουμε τη βιομηχανία να αποχωρήσει από την Ευρώπη. Επίσης θεώρησα ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουμε το, το ίδιο το MSR γιατί όπως ξέρετε το σύστημα ανταλλαγών εκπομπών, το ETS, αφορούσε αυτούς που θέλουν αυτά τα όρια, αλλά δεν είναι σκόπιμο να πιέσουμε ε, με βάση το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς. Θα πρέπει επίσης να δούμε και το θέμα της ε, διαφάνειας. Στους διαγωνισμούς δεν υπήρχε απόλυτη διαφάνεια. Και αυτό που μας ε, ενδιαφέρει είναι να ακολουθούμε τη διαδικασία ε, πλειοδότησης με βάση την ανάθεση έργων. Με ενδιαφέρει λοιπόν να το δούμε το θέμα εξονυχιστικά, θα φτάσουμε σε προτάσεις συμβιβασμού και όπως είπα θέλουμε να φτάσουμε σε μία πλειοψηφία διαφορετικά. Η Επιτροπή θα είναι πιο αδύναμη και εάν ε, αποτύχουμε τότε η πίεση της Κομισιόν θα είναι πολύ ψηλότερη. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ντελάνγκε από το ΕΛΚ, η πρώτη Σε Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Είχα πολύ χρόνο να διαβάσω την έκθεσή του και πόσο μπορώ να πω σχεδόν τη γνωρίζω, τη έχω μάθει απ' έξω γιατί έχουμε δουλέψει εδώ και μήνες θα ήθελα να δούμε ορισμένα ζητήματα όπου συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Πάση περιπτώσει θα πρέπει να γίνει κάποια εργασία μεταξύ ομάδων. Όπως είπα και πριν από το ΕΛΚ θεωρούμε ότι δεν είναι θέσφατα όσα προτείνει το Συμβούλιο και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε μαχή για να δούμε για κατά πόσο μπορούμε να αλλάξουμε τα ελεύθερα όρια και τα ε, όρια μετά από δημοπράτηση. Να αλλάξουν δηλαδή οι ποσοστιαίες αναλογίες. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, υπάρχει ίσως μία λίγο διαφορετική ε, στάση. Δηλαδή, εκεί αναφέρεται ε, ότι θα πρέπει να δούμε το ζήτημα μόνο εάν πραγματικά ανακύψει το θέμα των ορίων των ελευθέρων, των ανώτατων επιτρεπτών ορίων και των ορίων μετά από δημοπράτηση. Σε σχέση με τον κατάλογο διαρροής άνθρακα, παρόλο που το ε, κοιτάξαμε το θέμα ιεραρχικά και φαίνεται δελεαστικό, γιατί μιλάμε για καλύτερη στοχοθέτηση έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε και τα επιτρεπτά όρια καλύτερα. Όταν υπάρχει όμως οριοθέτηση θα πρέπει να δούμε, ε, να λάβουμε υπόψη ότι τα στοιχεία δεν είναι πάντα αξιόπιστα, όμως υπάρχουν θετικά και αρνητικά τη στιγμή που γίνονται οριοθετήσεις. Γι' αυτό θα προτιμούσαμε να έχουμε τη διτή προσέγγιση ε, τη διαδική προσέγγιση της Κομισιόν σε σχέση με τη δημοπράτηση και τα ελεύθερα επιτρεπτά όρια θα πρέπει να έχουμε πιο ρεαλιστικά στοιχεία όταν μιλάμε για κατανομή σε σχέση με, το, με την αύξηση 10% όπως προτείνει ο εισηγητής σε σχέση με την οριοθέτηση με το benchmarking θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούμε και το θέμα των εκπομπών οι οποίες είναι αναπόφευκτες και να έχουμε μία μείωση σε ορισμένες κατηγορίες κάτω από το 0,3% που πρότεινε ο εισηγητής. Βλέπω ότι κοιτάτε το ρολόι σας, Πρόεδρε. Και γι' αυτό το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι ο συντελεστής ε, διόρθωσης ίσως να μην ξεκινήσει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη στοχοθέτηση. Ο ε, ε, χρησιμοποιεί τη λέξη may αντί για should. Νομίζω ότι θα πρέπει όμως να αφήσουμε εν μέρη μία μικρή ευελιξία στα κράτη-μέλη. Αν θέλει ο εισηγητής μπορούμε να το συζητήσουμε. Παραμένω εδώ. Και ένα τελευταίο ζήτημα, όχι βέβαια τελευταίο, δεν θέλουμε να υπερφορτώσουμε τον εισηγητή με τροπολογίες, απλώς να δούμε τα βασικά ζητήματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τα κατόφλια έτσι ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία. Δεν μίλησα για το Ταμείο Εξυγχρονισμού και το Ταμείο Καινοτομιών, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, θα συνεργαστούμε στενά για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για την Επιτροπή Ήτρε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε ενώπιον μας το σαν Ιβο Μπελέτ. Όχι τώρα μετά εσύ, μετά τη συζήτηση. Ε, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ εξ ονόματος της Επιτροπής ΕΝΒΗ Περιβάλλοντος, πολύ σημαντικό. Ο κύριος Εντουάρ Μαχτά, σοσιαλιστής και δημοκράτης και σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ και τον κύριο Φέντερ, λέει τον εισηγητή. Βεβαίως, κάθε φορά ε, ε μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά της έρευνας και ο ίδιος ε, με πάρα πολύ μεγάλη διαφάνεια και ανοιχτό πνεύμα συνεργαζόταν πάντα μαζί μας και χαίρομαι γι' αυτό. Κοιτάξτε, εγώ θα επικεντρωθώ σε τρία πράγματα, τα θετικά, τα αρνητικά και τις ελλείψεις, κατά την άποψή μας. Ποια είναι τα θετικά. Βεβαίως, έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε ε, ότι πάμε σε πιο φιλόδοξους στόχους, 75% για 50% προκήρυξης σε σχέση με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει οι ποσοστώσεις να έχουν κάποιο χρηματικό αντίτυπο και να μην είναι ε, οι άδειε δωρεάν. Είναι προσωρινό αυτό το μέτρο. Ε, δεν μας ικανοποιεί η πρόταση. Ε, θα πρέπει επίσης να βελτιώνεται το reporting και να αυξάνεται η διαφάνεια. Τα είπε όλα αυτά είναι ωραία και καλά. Και μια άλλη ενδιαφέρουσα ιδέα για το αποθεματικό, ε, το σημείο 12, ε, για το, τα νέα εισερχόμενα, το, η τροπολογία 12 ήταν, η τροπολογία 29 για τους κλιματικούς στόχους μετά τη Συμφωνία των Παρισίων όλα αυτά είναι πολύ καλές ιδέες και είναι τα θετικά. Έρχομαι τώρα στα αρνητικά. Μας λυπεί το γεγονός ότι έχουν φύγει τα κοινωνικά στοιχεία, η ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων. Υπάρχουν χώρες μεταβατικές και υπάρχει ένα ταμείο ε, ε, μετάβασης. Δεν μπορούμε ως διαμαγείας να βγάλουμε τις οικονομίες και την παραγωγή από τον άνθρακα, να τον εγκαταλείψουμε τελείως. Ε, για τη διακυβέρνηση, το άρθρο 10 δεν θα πρέπει μόνο να βασιστούμε σε οργανικά στοιχεία. Η πολιτική κατά της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να είναι μόνο στα χέρια τραπεζιτών. Εμείς ως συνομοθέτες δεν θα πρέπει να βάζουμε κριτήρια επιλεξιμότητας πέρα από την απλή αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τώρα, στη σταδιακή προσέγγιση κατά τμήματα και τους τομείς από που κινδυνεύουν να φύγουν οι βιομηχανίες, διαρροή άνθρακα δηλαδή και το benchmarking, ε, δεν έχουμε ε, κοινοποίηση ενημέρωσης, παραμένουμε σε επίπεδα του 2008 και μείωση αυτόματη 0,3%. Δεν ξέρουμε αμφισβητούμε αν είναι αυτό η σωστή προσέγγιση, είναι προσυζήτηση. Και επίση δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις ε, δωρεάν ποσοστώσει και τη μεταφορά του τρίτου πακέτου ενέργειας. Αυτό ήταν ο δεύτερος πυλώνας. Έρχομαι στο τρίτο τώρα της ελλείψη. Δεν λέμε τίποτα για τον ε, συντελεστή γραμμικής ε, μείωση στο 2,2% ετησίω δεν μας φέρνει στο στόχο το 2050 ούτε γίνεται σεβαστό το 1,5 βαθμό Κελσίου που είχε βάλει η COP21. Ε, έχει κάπως εξειδανικευθεί η εικόνα η διεθνής. Ακόμα δεν είναι ο ανταγωνισμός θεμητός ή ε, ίσως ούτε θα γίνει στην τέταρτη φάση. Και γι' αυτό το λόγο τα γνωρίζετε από την αρχή θεωρώ ε, να έχουμε ευρύτερη προσέγγιση, όχι μόνο τις δωρεάν ποσοστώσεις, γιατί εάν προσπαθούμε να συμβιβάσουμε τα συμβιβαστά, θα είμαστε σε αδιέξοδο. Δεν θα κερδίσουν όλοι, θα χάσουν όλοι. Και δεν θα γίνουν ε, σεβαστοί οι στόχοι και οι δεσμεύσεις μας. Και τέλος, Ήδη από τη μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να δούμε πώς θα εγκαταλειφθεί αυτός ο μηχανισμός των δωρεάν ποσοστώσεων, να είναι πιο ικανοποιητική η ρύθμιση και να υπάρχει ίσως και θεμητός ανταγωνισμός και των διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας ε, στο ιστορικό τους, αλλά και μεταξύ τους διακλαδικά. Γιατί οπωσδήποτε αυτό το θέμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και δεν τελειώνει εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Χένκελ, αντιπρόεδρος, εκ μέρους της ομάδος ΙΣΕΡ και σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να έχουμε υπόψη ότι έχει ένα στόχο το ETS. Όμως υπάρχουν και άλλοι στόχοι, όπως για παράδειγμα να διατηρηθεί ή να ε, αυξηθεί η επανεκβιομηχάνηση τάξη του 30% και εμπλοκή για τις μικρές χώρες. Και δεν έχουμε μόνο να ανησυχούμε για τη διαρροή του άνθρακα, αλλά και για τη διαρροή θέσεων εργασία. Και αν υπάρχει μια επιτροπή στο Κοινοβούλιο που να διώκει τους στόχους, αυτή θα πρέπει να είναι η δική μα επιτροπή. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το λόγο σύστημα δεν είναι ικανοποιητικό. 45% των εκπομπών, α μην ξεχνάμε, καλύπτονται από το ETS, όχι όμως το 55%. Και έχουμε και το πρόβλημα της ε, ε, μη συμπερίληψης της ε, των μεταφορών. Θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες, σας αναφέρω συντομία ορισμένες. Πρώτον, θέλουμε αύξηση των των δωρεάν δικαιωμάτων. Επίσης, πρέπει να αυξηθεί το όριο, πρέπει να τα κατοπτρίζουν αυτά τα όρια την πραγματική βιομηχανική δραστηριότητα και αν υπάρχει μη εκμετάλλευση του 2%, μη κατανομή, αυτό ε, μπορεί να οφείλεται στις παραχωρήσεις. Θα πρέπει επίσης να επικαιροποιούνται τα benchmark αν υπάρχει πραγματική τεχνολογική πρόοδος. Επίσης θα πρέπει η μεθοδολογία για να πω στο κατάλογο διαρροής άνθρακα κάποιες θα πρέπει αυτό να βασίζεται σε ποιοτική ανάλυση. Την προσέγγιση αυτή τη θεματική tiered approach δεν τη δέχομαι. Δύσκολο είναι να ορίσουμε cost pass-through capability κατά αξιόπιστο τρόπο. Επίσης, θα πρέπει να αντισταθμίζεται πλήρως το έμεσο κόστος το Ταμείο Καινοτομίας πρέπει να παραμείνει ως έχει και να μην αυξηθεί. Τέλος, αυτά τα δωρεάν δικαιώματα να δίνονται μόνο σε όσους δίνουν δεδομένα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα ευνοήσει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά τις μεγάλες εταιρείε που μπορούν να τα συλλέγουν αυτά τα δεδομένα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εκ των Πρασίνων, ο κ. Ταλούντε. Η είναι ο σκιός Να σας καλωσορίσουμε γιατί αντικαθιστάτε και τον κύριο Έριξον που είναι πλέον μέλος της κυβέρνησης. Η Τροπή Ήτρε είναι γνωστή ως εξαγωγέας υπουργών στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Συνηθισμένο για μας λοιπόν. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Φρέντικ Φέντερλε για την πρότασή του που πιστεύω ότι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι μια βελτιωμένη έκδοση σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν, ιδίω ό,τι αφορά τη στοχευμένη προσέγγιση για τη διανομή των δωρεάν δικαιωμάτων ή την πρόταση για μεγαλύτερη διαφάνεια του συστήματος. Ευπρόσδεκτες όλες αυτές τις προτάσεις. Ωστόσο, θα ήθελα να υποστηρίξω πως η πρόταση της ΙΤ εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς φιλόδοξη και μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο για να είναι κατάλληλο για το σκόπο που έχει να επιτελέσει το ETS. Η πρόταση όσο έχει αυτή τη στιγμή δεν συνάδει ούτε με το στόχο του 2% ούτε με τις, ε, τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Αν αναβάλουμε τη λήψη των φιλόδοξων αποφάσεων τώρα και αν δεν δράσουν φασιστικότητα τώρα και οι επιχειρήσεις αλλά και οι πολίτες στην Ευρώπη τελικά θα πρέπει να καταβάλουν υψηλότερο τίμημα και πιο οδυνηρό τίμημα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία στο πλαίσιο του ETS που αντιβαίνουν στην όλη λογική του συστήματος. Αντιστάθμιση του έμεσου κόστους άνθρακα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, ιδίως που καταναλώνουν πολύ ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι διαστρεβλώνουμε την αγορά και αυτοί που ρηπαίνουν επιβραβεύονται. Ένα άλλο παράδειγμα, το άρθρο 10C που χρησιμοποιείται για αύξηση του, της, ε, του κύκλου ζωής ε, του ε, άνθρακα και των πολύ ρηπαινόντων σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και γεννητριών. Πρέπει οι χώρες με χαμηλό εισόδημα να μπορέσουν να εξυγχρονίσουν τον τομέα του ρεύματος και χρειάζονται τη βοήθεια. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού είναι κατάλληλο Εγώ θα έλεγα μέχρι το 2020 να καταργηθεί σταδιακά το 10 και να αυξηθεί η συμμετοχή του Ταμείου Εξαγωνισμού που είναι το πλέον κατάλληλο γιατί απευθύνεται σε όλους, ε, στις χώρες στους ίδιους ακριβώς τομείς. Είπα επίσης ότι είμαι υπέρ της πρότασης του εισηγητή για την ε, προσέγγιση αυτή που λέγεται tiered approach ό,τι αφορά την κατανομή των δωρεάν δικαιωμάτων. Επίσης θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την απαλλαγή από τον άνθρακα. Γι' αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι στην προσέγγισή μας. Η αρχή ορυπαίνων πληρώνει πρέπει να ενισχυθεί. Κανείς το δεν θα πρέπει να παίρνει βέβαια 100% δωρεάν δικαιώματα. Όλοι πρέπει να ξεκινήσουμε να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο Παρίσι. Θα πρέπει να σταματήσουμε να επιδοτούμε το ορυκτά καύσιμα και να χρησιμοποιούμε την δύναμη της αγοράς ώστε η Ευρώπη να γίνει ε, μια οικολογική καθαρή οικονομία που θα βασίζεται κάτω σε ανανεώσιμε πηγές ενέργεια. Ε, Τέλο, το ETS πρέπει να είναι πιο φιλόδοξο και πρέπει να εκπέμψουμε τα σωστά μηνύματα προ του ε, επενδυτές και στη βιομηχανία. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή πρόταση ω Ήτρε. Θα συνεργαστούμε με τον ΣΥΤΡΕ και του υπόλοιπου κοιόδη για αυτό το θέμα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιλικιώτης από την Αρχικά και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον συνάδελφο Φέντερ Λέι, για τη δουλειά που έκανε, για τι ενημερωτικέ συναντήσει που διοργάνωσε, αλλά και την προθυμία βεβαίω να συνεργαστεί με όλε τι πολιτικέ ομάδε ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για την ομάδα μα, την ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, πρωταρχικό στόχο τη αναθεώρηση του συστήματο πρέπει να είναι η μείωση των εκπομπών για προστασία του περιβάλλοντο και ενίσχυση τη ποιότητα ζωή των ανθρώπων και εμεί θεωρούμε ότι προ αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να υπάρξουν αυστηρότερα μέτρα για του μεγαλύτερου ρηπαντέ. Όσον αφορά τα δωρεά δικαιώματα σε τομεί που κινδυνεύουν, τονίζουμε πω πρέπει να δίνονται με αναβαθμίσει και στοχευμένα με αυστηρά κριτήρια ώστε να υποφελούνται οι βιομηχανίε που έχουν πραγματική ανάγκη. Εξίσου σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν από το σύστημα του μικρού ρηπαντέ. Όσον αφορά τέτοιε κρατικέ ενισχύσει, είναι σημαντικό για μα να συνεχίσουν να υπάρχουν ώστε να στηρίζονται οι μικρέ βιομηχανίε, διασφαλίζοντα έτσι ταυτόχρονα και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Ιδιαίτερα εν μέσω τη οικονομική κρίση πρέπει να στηρίξουμε τι μικρέ βιομηχανίε. Στα κράτη ιδιαίτερα που έχουν πληγεί περισσότερο από τι πολιτικέ λιτότητε, από τα μνημόνια, να φέρω μόνο ένα παράδειγμα, ε, και το παράδειγμα είναι τα κεραμοποιία, τα τσιμετροπία στην Κύπρο. Μιλούμε για μεσαίες, επιχειρήσει, επιχειρήσεις, καθώς και άλλες μικρές βιομηχανίες στον Νότο, η οποία ο Νότος σήμερα, ο Νότος της Ευρώπης, βρίσκεται σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Έτσι βεβαίω προστατεύοντας αυτές τις μικρές βιομηχανίες, προστατεύουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά ε, προστατεύουμε ταυτόχρονα και το περιβάλλον. Ε, είναι στη βάση αυτών των θέσεων και απόψεων μας που καταθέσαμε τροπολογίες ευελπιστούμε ότι εμείς ε, θα αποτρέψουμε τη δημιουργία ενός συστήματος εκπομπών που θα βοηθά τις μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες είναι και κύριες υπέτειες αυτές οι μεγάλες βιομηχανίε, των κλιματικών αλλαγών στο τέλος της ημέρας να αξιοποιήσουν αυτό το σύστημα για να αυξάνουν τα κέρδη τους σε βάρος των συμφερόντων ολόκληρης της κοινωνίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι, σας ευχαριστώ όλους και τον ε, εισηγητή και τους σκιώδης. Και τώρα πάμε στους άλλους ομιλητές. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να θέσω υπόψη της ε, Επιτροπής και θα καταθέσω και σχετικές τροπολογίες το ζήτημα της απαλλαγής από την υποχρέωση της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα κράτη-μέλη με κατακεφαλή ΑΕΠ χαμηλότερο του 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έτος αναφορά το 2013 απαλλάσσονται από την υποχρέωση της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων. Η Ελλάδα, παρότι ξεπερνούσε ελαφρώς αυτό το κριτήριο, γιατί είχε κατακεφαλή εισόδημα το 2013 62%, εν τούτης πληρεί αυτό το κριτήριο για το 2014, καθότι το ποσοστό είναι 59,7%. Το ποσοστό ήδη έχει πέσει λόγω των μνημονίων, των μέτρων λιτότητας, δημοσιονομικής προσαρμογής, της φτωχοποίησης της χώρας, έχει πέσει για το 2015 στο 56,5% του ΑΕΠ. Και δυστυχώς φοβάμαι ότι και για το 2016 θα είναι τα πράγματα χειρότερα. Επομένως, αυτή τη στιγμή, <clears throat> από τις γειτονικές χώρες στην Ελλάδα, μόνο η Ιταλία δεν έχει μπει στην εξαίρεση. Οι άλλες χώρες, είτε είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν εξαίρεση, είτε είναι τρίτες χώρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται στρέβλωση στον ανταγωνισμό και να αποτυπώνεται κυρίως σε αυξημένες ελληνικές εισαγωγές ρεύματος, με αποτέλεσμα να απειλείται η βιωσιμότητα της ΔΕΗ, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Να επισημάνω ότι πλέον ε, υπάρχουν αυξημένες τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα, ότι υπάρχει αύξηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα και ότι υπάρχει απώλεια της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιριών. Ήδη στις 27 Μαΐου έχω υποβάλει μια σχετική ερώτηση στην Κομισιόν και νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει δεκτή ή να γίνουν δεκτές δύο τροπολογίες τις οποίες θα καταθέσουμε εντός της προθεσμίας, αύριο, ούτω ώστε να μπορεί και η Ελλάδα να, παρότι δεν είχε το κριτήριο του έτους αναφοράς το 2013, αλλά το πληρεί το 2014, δηλαδή έχει χαμηλότερο του 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορεί να ενταχθεί σε αυτή την εξαίρεση, ούτως ώστε να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να απαλλαγεί από την υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αέριων. Αυτό πολύ περισσότερο σε μια χώρα όπου χρησιμοποιείται κυρίως ο λιγνίτης αυτή τη στιγμή. Εάν γίνουν δεκτέ αυτέ οι δύο τροπολογίε, γιατί θα κάνω αντίστοιχη τροπολογία και για το Ταμείο Εξυγχρονισμού που υπάρχει και καινοτομία, τότε θα μπορέσει να στηριχθεί η πατρίδα μου σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που χρειάζεται να αποκτήσει μια ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία λόγω χαμηλών τιμών ε, ενέργειας. Αυτά είναι τα δύο σημεία που θέτω υπόψη και στον εισηγητή, τον οποίο ευχαριστώ ε, για την δουλειά που έχει κάνει και βεβαίως τους υπόλοιπους συναδέλφους, ενημερώνοντας ότι θα καταθέσω αυτές τις δύο τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much, ε, Mr. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπεθ. ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πάει στη σωστή κατεύθυνση η δουλειά και συμφωνώ και με τον συνάδελφο Μαρτά. Θα πρέπει να ενισχυθεί το σχέδιο έκθεσης, να βελτιωθεί και να μπουν κάποια στοιχεία που μας λείπουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το κοινωνικό επίπεδο, όπως ακούστηκε και προηγουμένως. Ε, θα ήθελα από πλευράς μου να επιμείνω στην ανάγκη αποζημίωσης η αντιστάθμιση του άμεσου κόστους από την Ευρώπη για εκείνου του τομείς που εκτίθενται περισσότερο στη διαρροή άνθρακα. Το 2015 πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ πήγανε σε αποζημίωση ε, ε, έμεσου κόστους. Αυτό είναι μεγάλη δαπάνη και εξαρτάται από τη δυνατότητα τη δημοσιονομική της κάθε χώρας, του κάθε κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά και ε, οθεί σε αθέμητο ανταγωνισμό την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Για να εναρμονιστεί καλύτερα και να ρυθμίζεται η αγορά, τι προτείνουμε εμεί και θα το κάνω και εγώ με τροπολογία. Να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο αποζημίωση των εμέσων ε, ε, δαπανών τουλάχιστον 2% των δικαιωμάτων από το 2021 στο 2030. Από την άλλη θα πρέπει να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο για εκείνους τους τομείς που από τις διαδικασίες παραγωγής δεν μπορούν να έχουν αντίστοιχα μέτρα. Ας πούμε υπάρχει συμπαραγωγή ενέργειας και ε, θερμοκοτήτας υψηλή ποιότητα που δεν θα πρέπει να τα πληρώσει τα σπασμένα. Χρειάζεται βάθυνση σε κάποια στιγμή και σε κάποια άλλα βελτίωση ή πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τα σχόλιά σας. Ο κύριος Νταν Νίκα. Θα ήθελα να αρχίσω με ένα γενικό σχόλιο. Υπάρχουν πολλές ανακρίβειες στο έγγραφο της Επιτροπής και ελλείψεις. Δεν έγινε διαβούλευση, δεν υπήρξε διαφάνεια όπως διαπίστωσε. Εγώ έστειλα μία επιστολή για να ρωτήσω ε, ποια θα πρέπει να είναι τα benchmarks για την ενεργειακή απόδοση και τους είπα ότι θέλω να μου πείτε ε, ποιες είναι οι χώρες που έχουν τη ε, μεγαλύτερη απόδοση. Δεν μου δόθηκε καμία ε, απάντηση εκτός για τα έτη 2007-2008. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που είπαν ε, οι κύριοι Φέντερλε και Μαρτέν ήταν πολύ σωστά. Δηλαδή, δυστυχώς, ε, δεν υπάρχει διαφάνεια στην ε, παράδοση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει με, αυτή τη, με αυτό το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο να αυξηθεί η τιμή της ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ε, ότι έχουμε 60 ε, εκατομμύρια τα οποία θα πρέπει να διατεθούν και θα πρέπει να είμαστε και ανταγωνιστικοί και να ε, βρούμε νέες θέσεις εργασίας. Μιλάμε για μια αύξηση του κόστους κατά 20%. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Απολύτως απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας ούτε για τους ιδιώτες ούτε για τις βιομηχανίες. Ε, το phase out το βλέπει με μεγάλη ελαφρύτητα η Κομισιόν. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη χώρα μου θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες και στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της ε, αύξησης της ε, τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό για τα νοικοκυριά. Καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στα τιμολόγια της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Θα πρέπει να υπάρξουν καινοτομίες, αλλά δεν μπορεί να ε, καταβάλουν το αντίτιμο οι οικογένειες και τα παιδιά τους. Πολλά υπόθηκαν στον ε, τεχνικό τομέα. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, αλλά δεν νομίζω ότι από τεχνικής πλευράς μπορούν να επιβληθούν μέτρα τα οποία ε, αποτελούν μία γραμμική διόρθωση. Υπάρχουν πολλές ε, καμπύλες και σκαμπαναβάσματα στις τιμές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν μπορούμε παρά να δεχτούμε τα πραγματικά στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν να αναγνωρίσει τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου και αν δεν είμαστε αλληλέγγυοι όλοι τότε θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ δυσάρεστες συνέπειες ως προς την τιμολόγηση. Η κυρία Γκροστέτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία του. Πρόκειται για ένα θέμα ύψης της σημασίας για την Ευρώπη. Όλοι θεωρούμε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά θα πρέπει να βρούμε μέτρα διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας. Ε, με βάση έναν ε, ε, ανταγωνισμό, αμήλικτο ανταγωνισμό παγκοσμίω. Μιλάμε βεβαίως για διαρροή άνθρακα και διαρροή επενδύσεων. Οι προδιαγραφές μας είναι υψηλές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι δικές μας βιομηχανίες θα πρέπει να παράγουν αλλού με χαμηλότερες προδιαγραφές. Δεν ε, δέχομαι ότι θα πρέπει να διαγραφεί αυτή η δυνατότητα ε, αποτίμησης της ε, διαρροής άνθρακα με βάση ποιοτικές ε, μελέτες. Θα πρέπει να βρούμε μία εξισορρόπηση για να έχουμε μία τιμολόγηση όπου θα μπορούν να γίνουν σωστές επενδύσεις και να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τις ποσοστός που έχει στη διάθεσή του. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε το περίφημο 57% που αφορά τα δικαιώματα ε, με βάση το, τους διαγωνισμούς και τις, ε, τα ελεύθερα δικαιώματα, τα δωρεάν δικαιώματα που είναι το υπόλοιπο και δεν μπορούμε να αποδίδουμε πολύ υψηλέ ποσοστώσει σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους που απέτυχε το ETS μέχρι τώρα. Θα πρέπει να έχουμε, μάλλον αυτά τα δεδομένα υπάρχουν, γι' αυτό θα πρέπει να κατανεμηθούν αυτές οι ποσοστώσεις ανάλογα με το επίπεδο παραγωγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. για να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος βεβαίω. Ο κύριος Κολίτσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μερικά σχόλια να κάνω κι εγώ από την πλευρά μου. Η αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Μπορεί να είναι σωστή, αλλά να μην υπερβάλλουμε κιόλα. Γιατί μετά θα έχουμε ένα καθαρό περιβάλλον και από δουλειά τίποτα. Σας είπα το γυαλί ε, είναι ε, υλικό που χρησιμοποιείται και για τις ε, συσκευασίες. Αυτό μπορεί να μεταφερθεί κάπου, αλλά όχι σε μεγάλη απόσταση, διότι είναι ακριβό και κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτές τις εργασίες να σηκωθούν να φύγουν. Βεβαίως να μειωθεί η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, δεν λέω, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και τι κάνουμε για να κρατάμε τις δουλειές στην Ευρώπη από ποιο ταμείο, δηλαδή θα αποζημιώσουμε τους ανέργους που θα προκύψουν και τι θα κάνουμε για αυτούς, για να μπορεί στην πράξη να λειτουργεί αυτό το σύστημα, όχι να λέμε μόνο 2%. Εντάξει, και από εκεί και πέρα σε ορισμένες χώρες Έχουμε θέρμαση με κεντρική θέρμαση που στέλνουμε σε διάφορες συνοικίες ε, και αυτά θα πρέπει να μπορούν να τα χρησιμοποιούν και εταιρείε. Αν δεν έχουμε εταιρείε να τα χρησιμοποιούν θα προκύπτει πολύ περισσότερη ρήπανση από αυτό το είδος της θέρμασης Δεν μπορούν, υπάρχουν κλάδοι της βιομηχανίας που εκπέμπουν ρήπους. Σε ό,τι αφορά τους διάφορους συντελεστές και τα ποσοστά θα πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι τα οριστικά. Φυσικά θα κάνω και εγώ τροπολογίες ε, σχετικές ε, για το θέμα αυτό της κεντρικής θέρμας από Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και καιρό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι έχω επιφυλάξεις για το σύστημα ETS εμπορίε εκπομπών και από το δρόμο που έχει πάρει και τις εξελίξεις. Ε, είναι μια αγορά που δημιουργήθηκε τεχνητά. Δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι στη θέση του κυρίου Φέντερλε, δεν το ζηλεύω. Είναι πολύ περίπλοκη η δουλειά αυτή και να βγάλεις κάτι το ισορροπημένο και λογικό. Αν θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών, λοιπόν, ETS, θα πρέπει πραγματικά να ξέρουμε πώς έχουν οι προϋποθέσεις στα διάφορα κράτη-μέλη και να τις λαμβάνουμε υπόψη μας, την κάθε πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει να κάνουμε και άλλη ζημιά στη βιομηχανία μας, εάν δεν είναι σωστά μελετημένο το σύστημα ε, θα πάθουμε ζημιά. Το άρθρο 10C και 10D είναι πολύ προβληματικό από τη σκοπιά πολλών κρατών μελών και δεν μιλώ μόνο για τις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η έκθεση λοιπόν με τη μορφή που έχει ε, σήμερα νομίζω δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνος. Δεν ισχύουν αυτά που λέει στο 10C και στο 10D. 10 εκατομμύρια νομίζω θα πρέπει να είναι το όριο εκεί και να μην καταργηθεί. Στο 10D το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιτίθεται με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και έχουμε πρόβλημα. Θα πρέπει στα κράτη-μέλη να αποφασίζεται η ε, ε, κάστοτε ε, ρύθμιση, γιατί οι χώρες ξέρουν καλύτερα και την κατάσταση που επικρατεί εκεί και τις βιομηχανίες τους. Έχουμε πάρει άλλη κατεύθυνση όμως. Ο, ο εισηγητής προτείνει κάτι πολύ περίπλοκο που δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Οπότε, θα κάνουμε και εμείς τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Και ελπίζω να ε, καταλήξουμε σε ένα καλό κείμενο με ισορροπία και που να σέβεται όλες τις πλευρές και όλες τις ιδιάζουσες συνθήκες για να βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν. Ο κύριος Γκάια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τους ηγητές, τους κοιότητες και τον εισηγητή τον ίδιο. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η δουλειά, πάρα πολύ υπεύθυνη από πλευρά της Επιτροπής μας και θα πρέπει με την ησυχία μας ε, να εμβαθύνουμε ε, στη συζήτηση για να βάλουμε τα σωστά θεμέλια. Εγώ έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Τι θέλουμε πολιτικά να επιτύχουμε. Θέλουμε μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό πρότεινε η διάσκεψη των Παρισίων. Ή θέλουμε να δώσουμε ένα ε, μήνυμα υψηλών τιμών. Και αν είναι υψηλέ οι τιμέ, δεν θα οδηγήσει αυτό αναγκαστικά στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να βάλουμε και άλλους τομείς οπωσδήποτε στο ETS, αν θέλουμε να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Ο συνάδελφος Βεν Λάγκ θα κάνει μια τροπολογία για να μπει και η ναυτιλία. Οι ε, θαλασσίες μεταφορές εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Από εκεί και μόνο θα μειωθεί ε, το διοξίδιο του άνθρακα χωρίς να είναι υψηλές οι τιμές για τη βιομηχανία. Γιατί αρχή του ο πληρώνει τελικά ε, αντιτίθεται σε ένα στόχο της Ένωσης. Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι θα συμφωνούσα με τον κύριο Χιάνκελ στη ζωή μου πολιτικά, το είδαμε και αυτό, ε, θα πρέπει να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας και 20% της παραγωγής ε, πλούτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βιομηχανική παραγωγή. Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα ε, των κρατών μελών κλάσμα που δεν φτάνει στο 20%. Η Γερμανία, η πατρίδα μου, ευτυχώς είναι εκεί και θέλω να παραμείνει και να μην χάσουμε αυτό το βιομηχανικό πλούτο. Και δεν είναι καθόλου old economy. Προηγουμένω είδαμε πόσο καινούριο είναι αυτό ο κλάδο και πόσο σύγχρονο. Και θα πρέπει ε, στη νέα περίοδο του ETS να ληφθούν όλα αυτά υπόψη και να τα δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Είμαι ακράδαντα πεπισμένο ότι η γραμμή που λέει το 10% των πιο αποτελεσματικών κλάδων ε, θα πρέπει να μείνει εκτός ε, πιστοποιητικών πρέπει να διατηρηθεί έχει απόλυτο δίκιο ο συντονιστή μου, ο Νταν Νίκα, γιατί μέχρι τώρα δεν ξέρουμε καθόλου, δεν έχουμε ιδέα πού κατεβάζει αυτά τα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πού τα βρίσκει. Μία είναι η ερμηνεία που είναι ε, απλά μαθηματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαρτίζεται από καλού υπαλλήλου και γενναίου, το λέω χωρί καμία ηρωνία, και ε, του είπαν από το Συμβούλιο ε, να είναι 75% προς 43% και κάνουν απλή αριθμητική και βγάζουν κάποιους στόχους. Ε, αυτά λοιπόν είναι και τέλος έρχεται και ένα benchmark. Πλην όμως το χαζό είναι ότι σε ορισμένες ε, βιομηχανίες όπως τη τσιμεντοβιομηχανία, τη χαλιβουργία δεν γίνεται αυτό για λόγους των νόμων της φυσικής γιατί το Κοινοβούλιο, ακόμα το Ευρωπαϊκό, τη φυσική δεν μπορεί να την καταργήσει και θα πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη. Αν θέλουμε λοιπόν το 10% των πιο αποτελεσματικών εργοστασίων να εξαιρούνται από το χάος αυτό των ε, πιστοποιητικών, να παραμείνει έτσι. Να το εξασφαλίσουμε και γι' αυτό συμφωνώ με την ιδέα για το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς. Εμείς το δημιουργήσαμε αυτό για να στείλουμε ένα μήνυμα για τις τιμές, για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Σωστό ήταν τότε όταν το κάναμε. Αλλά επειδή είχαμε την κρίση κατέρευσαν οι τιμές και αν θέλουμε κάποια στιγμή να την ξεπεράσουμε, όταν με το καλό περάσει η κρίση, καλό θα ήταν να εξαιρεθούν αυτοί οι κλάδοι ε, της βιομηχανίας. Πιστεύω, όχι δεν πιστεύω, γνωρίζω ότι στη Γερμανία ευτυχώς έχουμε υψηλή απασχόληση και υψηλή βιομηχανική απασχόληση. Εγώ είμαι από το Ρούργκεμπιτ, από την περιοχή του Ρούρ και αυτά δεν ισχύουν. Είμαστε από τις πόλεις με τη μεγαλύτερη ενεργεία στη Γερμανία και δεν μπορώ να συμφωνήσω με ρύθμιση που θα μου λένε τα συνδικάτα ότι θα έχουμε και άλλους ανέργους στη βιομηχανία στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αγγέλ Κανίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ζητώ συγγνώμη που μόλις έφτασα και δεν κατάφερα να παρακολουθήσω τη συζήτηση. Δύο-τρία σχόλια από πλευρά μου. Α, φτάσατε πάνω στην ώρα, λέει ο Πρόεδρος, δεν έχετε καθυστερήσει καθόλου. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε δύο στόχους. Το πρώτο είναι ο φιλόδοξος στόχος για την προστασία του κλίματος 40% μέχρι το 2030 και έχουμε και διεθνείς ε, δεσμεύσεις, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και άλλο στόχος, το είπα και συνάδελφοι, να μην μας φύγουν οι θέσεις εργασίας από την Ευρώπη. Να διατηρηθεί και να ενισχυθεί μάλιστα η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και αυτά τα δύο να μπορέσουν να συγκεραστούν. Αυτό είναι το μέγα ζητούμενο τώρα. Τώρα, στο θέμα αυτό, ξέρετε ότι ε, είμαι από μια εκλογική περιφέρεια όπου Έχουμε χημική βιομηχανία, τσιμέντα, χαρτί, αυτοκίνητα, γυαλί και δεν συμμαζεύεται. Όλοι αυτοί οι κλάδοι θίγονται από το εμπόριο εκπομπών. Καταλαβαίνετε τι εκνευρισμό επικρατεί και βλέπω και τι τεράστιε προσπάθειε. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο κύριος Νίκα, κάποιο πρόβλημα έχει η ρουμανική διερμηνία. Τώρα είναι εντάξει. Οκ. It's okay. Can, can be helpful. Τώρα είναι εντάξει, ακούγεται. Good. No, no, no, it's okay, it's okay, it's perfectly okay. You, you should, you should follow it, everyone. Okay, βεβαίως, λοιπόν. Έλεγα λοιπόν ότι θίγονται διάφοροι κλάδοι και δυστυχώς, καθόλου δυστυχώς χαίρομαι που όλε αυτές οι βιομηχανίες είναι στην εκλογική ε, περιφέρεια, αλλά έχουν ανησυχήσει, έχουν θορυβηθεί και θέλουν να είναι αποτελεσματικοί, να κάνουν οικονομία ενέργειας, να μην εκπέμπουν, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια στιγμή ε, αγγίζουμε και τα τεχνολογικά ε, όρια να σφίξουμε ε, τη στρόφιγγα, αλλά υπάρχει και όριο. Να δούμε το ποσοστό των δωρεάν ε, δικαιωμάτων και των ε, ε, προκηρύξεων των δημοπρατήσεων, των πληστηριασμών, 75 και 43. Όλα αυτά είναι θεωρητικά και μαθηματικά. Εκεί θα πρέπει να το ξαναδούμε αν είναι σωστή αυτή η στόχη. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, διορθωτικοί συντελεστές ε, που δεν με βρίσκουν σύμφωνοι γιατί το θεωρώ άδικους. Επειδή έχει προχωρήσει η ώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες το benchmark, τα στοιχεία από το 2008 θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, να ενημερωθούν. Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση και αν δεν έχει βελτιωθεί ε, θα πρέπει να διατηρηθεί και ε, να μην γίνει πιο αυστηρό το μέτρο έτσι, κατά αποκοπή που να ισχύει για όλους. Θα κάνουμε τροπολογίες για να θα συζητήσουμε. Κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιες εκπομπές που έχουν ε, κάνουν με τη μέθοδο ε, παραγωγής. Δηλαδή υπάρχει ε, ένας κλάδος ή πολλοί κλάδοι της βιομηχανίας που δεν μπορούν να βελτιώσουν τις μεθόδους για να εκπέμπουν λιγότερα. Τι θα γίνει λοιπόν με το έμεσο κόστος και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Η εθνική λύση είναι καλή νομίζω για τα κράτη-μέλη να μπορούν να το αποφασίζουν. Αυτά και τελείωσα. Και ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ήταν δύο επί δύο, επειδή υπήρξε αυτή η διακοπή, χάρη στον Ντανίκα βέβαια. Πολύ δύσκολο το καθήκον του συντάκτης νομοδότης. Φαντάζομαι πιο δύσκολο είναι και το έργο του συναδέλφου εισηγητή από την Επιτροπή εβ Ιβο Μπέλετ. Αγαπητέ κύριε Μπέλετ, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να σας ακούσουμε, εφόσον είστε και ο υπεύθυνο, ε, όχι μόνο για την ε, λογαριασμό της Επιτροπής αλλά για όλη την... Ε, για Μα ξέρετε, όχι, είμαι ο εισηγητής από το ΕΛΚΑ απλά. Αν μου επιτρέπετε να κάνω λίγες παρατηρήσεις, ε, να ευχαριστήσω καταρχάς για τη φιλοξενία Ήμουν εισηγητής ε, για το φάκελο MSR και πράγματι είχαμε πολύ καλή συνεργασία οι δύο επιτροπές, ε, Ήτρε και Ένβη και θέλω να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η καλή συνεργασία με το Φρέντρικ για το φάκελο αυτό και στο μέλλον. Ο εισηγητής που δεν είμαι εγώ επαναλαμβάνω, συμφωνεί και αυτός. Νομίζω τώρα ότι συμφωνούμε πάνω σε πολλά κρίσιμα ε, ζητήματα, να σεβαστούμε τις δυνάμεις του Παρισιού, το στόχο για το 2030, ε, σημαντικά είναι τα, σημαντικό είναι το Ταμείο Καινοτομία, συμφωνούμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ώστε αυτό το μεγαλύτερο προπολογισμό. Συμφωνεί η Επιτροπή ΕΜΒΗ και ΙΤΡΕ ειδική μεταχείριση για τις ΜΜΕ και εδώ υπάρχει συνένεση νομίζω. Διαφωνούμε σε ό,τι αφορά την υλοποίηση κάποιων λεπτομεριών, αλλά θέλουμε να υπάρχει αυτή η καλή μεταρρύθμιση για τη, ε, μεταχείριση για τις ΜΜΕ. Μιλήσατε για τα μέτρα κατά της διαρροής άνθρακα. Φρέντρικ, δεν συμφωνούμε ε, και συμφωνώ με αυτό που είπε και η Έστερ ότι πραγματικά αυτή η προσέγγιση, η tiered approach, μας έχει μαγεύσει και το μελετήσαμε το θέμα πάρα πολύ διεξοδικά, κύριε Πρόεδρε, αλλά προτιμούμε την πρόταση της Κομισιόν τελικά. Είναι καλύτερη, πιστεύουμε. Εξυγχρονισμός, ταμείο εξυγχρονισμού. Διαφάνεια είναι πολύ σημαντική Επίσης ακούσαμε πολύ προσεκτικά τις παρατηρήσεις ε, αρκετών Ελλήνων συναδέλφων. Νομίζω έχουν έγκυρα επιχειρήματα και θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Επίσης ε, το έμεσο κόστος είναι κάτι που σχολίασαν πολλοί συνάδελφοι. Η δική μας θέση είναι όπως και αυτά που, που είπε η Έστερ Ντελάνγκε στην ΕΝΒ και, στην και στην Ήτρε, δηλαδή θέλουμε να υπάρχει πιο ισότιμο ε, πεδίο. Αλλά με ποιο τρόπο μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Τέλος. Η, παρέκ... η απόκληση, το deviation. Συγγνώμη, η αεροπορία aviation δεν αναφέρθηκε μάλλον. Ναι, όχι, δεν ανέβηκε. Τον συνάδελφο Ντάνκα να μας τον χαιρετήσετε, που είναι και ο εισηγητής. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρω ότι ήταν ε, έντονη η συζήτηση και στην Επιτροπή σας ο συνάδελφος Ντάνκαν να διορθώσω λοιπόν, είναι ο βασικό εισηγητή από το ομάδα ECR. E Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Διευθύντρια Πετέσκη από τη ΓΑΜΑ Κλίμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που συμμετείχατε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα συζήτηση. Μας ε, δώσατε πάρα πολλές πληροφορίες Ήδη βέβαια πρέπει να σας πω ότι απασχολούμεθα με αυτό το θέμα εδώ και καιρό ε, με τους κοιόδες εισηγητές έχουμε επαφές και προσπαθούμε να εξηγήσουμε την πρότασή μας καλύτερα. Ήρθε ο Επίτροπος, Γενικός ε, Διευθυντής, ε, πολλοί από εμάς. Ας εστιάσω λοιπόν εγώ μόνο σε κάποια ζητήματα, αυτά που συζητήθηκαν περισσότερο στη σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Όπως υπόθηκε στη συζήτηση, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ε, λεπτές πολιτικές επιλογές όταν θα σχεδιάσουμε για την επόμενη 20 ετία το ETS. Θέλω να το τονίσω αυτό. Και νομίζω να γνωρίστηκε και στη συζήτηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αφετηρία έλαβε τα συμπεράσματα του Οκτωβρίου 14 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτά μας καθοδηγούν. Και σε αυτά βασίσαμε την πρότασή μας. Έρχομαι σε λίγα ζητήματα που νομίζω ότι είναι και τα πλέον κρίσιμα. Διαρροή άνθρακα καταρχάς. Όπως γνωρίζετε, και το έχουμε πει πανελειμμένος το είπε και ο Επίτροπος, χαιρετίζουμε τη συζήτηση για τις διάφορες αυτές ε, απόψεις περί της προσέγγισης approach. Ήταν μία από τις αναλλακτικέ, αν θυμάστε καλά, που συζητήσαμε και στη μελέτη αντικτύπου που κάναμε. Θα συνεχίσουμε να ακούμε τη συζήτηση. Είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες. Βέβαια, Φαντάζομαι έχετε δει ότι η προτινόμενη προσέγγιση στο τη του ουσιαστικά οθετεί μία από τις προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη μελέτη αντικτύπου. Αναγνωρίζουμε όμως τη δυσκολία του όλου εγχειρήματο. Μια πιο στοχευμένη προσέγγιση βέβαια από την άλλη πλευρά Ίσως να μην ενεργοποιεί τόσο συχνά αυτό τον διορθωτικό συντελεστή, αλλά υπάρχουν και τα τεχνικά ζητήματα. Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε και στις μελλοντικέ συζητήσεις. Ποιοτική αξιολόγηση τώρα. Το αναφέρατε αρκετοί αφορά τομεί ε, ένταση ΜΜΕ. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων δηλαδή. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για μια ποιοτική αξιολόγηση για του τομεί εκείνου που βρίσκονται ε, στην κόψη, στο χείλος του ανώτατου, του κατώτατου όριου του κατφυλίου αυτού. Βέβαια θέλουμε να μειώσουμε το διοικητικό άχθος και η προσέγγιση του εισηγητή Σίγουρα το επιτυγχάνει αυτό. Και ίσως ε, επιτυγχάνεται και μεγαλύτερη διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Με την προσέγγιση αυτή όμως, νομίζω ότι πρέπει να στοχεύουμε παραλαμβάνω σε λιγότερη διαφά... γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια. Όσο πιο κοντά είμαστε στο κατόφλι. Η δωρεάν κατανομή, όπως ξέρετε, είναι μειωμένη και μειώνεται ακόμη περισσότερο. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει αυτός ο κατάλογος ε, διαρροής άνθρακα και να έχουμε τα σωστά benchmark. Έγινε αρκετή συζήτηση σήμερα για αυτό το θέμα. Γνωρίζετε φαντάζομαι, αλλά θα το εξηγήσω, θα προσπαθήσω τουλάχιστον για μια ακόμη φορά θα εξηγήσω ότι εμείς αναζητούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των κινήτρων και καινοτομία, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε στο μέλλον μια ανταγωνιστική βιομηχανία. Θέλουμε όμως ταυτόχρονα να έχουμε χαμηλό διοικητικό φόρτο και προβλεψιμότητα, επαρκή προβλεψιμότητα για τους τομείς. Στο σχέδιο γνωμοδότησης ε, λέγεται ότι θα πρέπει να μείνουν ε, οι ε, πρότυποι συντελεστές. Προτείνει επίσης έναν άλλο πρότυπο συντελεστή, standard rate, για να διασκεδαστούν σχέσεις ορισμένων κλάδων που μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες με το χαμηλότερο συντελεστή. Είμαστε ανοιχτοί να εξετάσουμε από κοινού αυτό το ενδεχόμενο, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το ίδιο το πλαίσιο. Έχω παραστεί σε πολλές συναντήσεις και άλλοι συναδελφοί μου και πρέπει να επισημάνω ότι φαίνεται να είναι κατανοητό ότι η πρόταση ε, της ε, Κομισιόν δεν λαμβάνει υπόψη πραγματικά δεδομένα αντίθετα. Όπως γνωρίζετε θα συλλέξουμε νέα δεδομένα παραγωγής και θα τα μελετήσουμε και θα τα διασταυρώσουμε για να δούμε ποιο είναι το αναπτυξιακό δυναμικό βάσει των ε, δεδομένων αυτών που θα συλλέξουμε σε σχέση με τον συντελεστή που εφαρμόζεται. Τον καταποκοπήν αυτό συντελεστή flat rate. Και πιστεύουμε ότι με τα δεδομένα θα αποδειχθεί ότι η τεχνολογική ανάπτυξη ήταν πολύ χαμηλότερη το 1%, 0,5% ε, είναι ο συντελεστή που θα εφαρμοστεί. Μπορώ να σα δώσω περισσότερε λεπτομέρειε ω εξήγηση, απλά ήθελα να σα δώσω έτσι μια πρώτη γεύση να καταλάβετε δηλαδή ότι δεν ακολουθούμε εδώ μια αμυγός γραφειοκρατική προσέγγιση, αλλά έχουμε επαφή και με την πραγματικότητα. Δύο λέξεις... Α, δεδομένα παραγωγής. Είπα ότι θα συλλέξουμε αυτά τα δεδομένα ε, και μάλιστα θα το κάνουμε δύο φορές στη διάρκεια της περίοδου, αλλά στην πρόταση μα ε, περιλαμβάνονται και προτάσεις ώστε να γίνεται πιο συχνά αυτή η παροχή των δεδομένων στη διάρκεια της περίοδου. Αυτό σχετίζεται με το κατόφλι του 10% που προτείνει ο εισηγητής. Θα ήθελα να είμαστε προσεκτικοί εδώ. Φυσικά και μας ενδιαφέρει να έχουμε μια καλύτερη ευθυγράμμιση. Θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη ότι αυτό συνεπάγεται και μεγάλο διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και για τα κράτη-μέλη και για την Κομισιόν. Άρα πρέπει να βρούμε τη σωστή λύση. Η Κομισιόν θεωρεί λοιπόν ότι καλό είναι να προηγηθεί μια ξεχωριστή μελέτη αντικτύπου και εν συνεχεία να καταλήξουμε σε μια προσέγγιση ε, σε ό,τι τη φάση εφαρμογής, αλλά να είναι συμμετρική προσέγγιση. Ο πρόεδρος δεν σας δια κόπτω, Να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω με ένα τελευταίο σχόλιο. Εφτά λεπτά μιλάτε όμως, λέει ο πρόεδρος. Ναι, αλλά με προκάλεσαν οι συνάδελφοί σας και νομίζω ότι καλό είναι να εξηγήσω λίγο καλύτερα την πρότασή μας. Λοιπόν, έχουμε και την κοινωνική διάσταση, το οποίο είναι ένα ζήτημα που αναφέρατε αρκετοί. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση των εσόδων των πληστηριασμών για τον δημιουργία δεξιοτήτων. Να σας πω ότι όμως έχουμε μελετήσει πάρα πολύ καλά όλες τις πτυχές. Ευχαριστώ. Θα το συζητήσουμε και με τον ε, εισηγητή μας το θέμα. Αν θέλετε, επειδή ήταν ευρύτατη η παρουσίαση, η εισήγηση της Επιτροπής, αν κάτι θέλετε να πείτε για μισό λεπτό, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να μου πει εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Growth και Energy πώς έχει ε, το θέμα. Δεν ε, είναι αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Κλίμα. Σας είπα για την αύξηση των τιμών κατά 20% και δεν έγινε κανένα σχόλιο για την ε, μελλοντική αύξηση των τιμών για τον καταναλωτή. Και αυτό είναι ντροπή. Άλλα σχόλια, συνάδελφοι. Μα η Γενική Διεύθυνση για το κλίμα είναι υπεύθυνη. Κάθε φορά που μιλώ με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας ή Growth ή Ανάπτυξης μου λένε κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Ήτρα και της Έμβη σε μας, στα κάθε μας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Ο εισηγητής μας έχει τον τελευταίο λόγο για σήμερα. Μα θα το συζητήσουμε φυσικά και στους επόμενους μήνες. Βλέπουμε ότι είναι ευρύτατη η συζήτηση και μπορούμε και να την εμβαθύνουμε πολύ. Ξέρω ότι από τεχνικής πλευράς ε, δεν έχουν γίνει όλα όσα θα ήταν δυνατά, δυνατό να γίνουν και θα ήθελα να σας μιλήσω για τη ρήτρα αναθεώρησης για το 2023, όπου μπορούμε ε, να προσαρμόσουμε τους στόχους στο νομοθετικό πλαίσιο και κάτι το οποίο με απασχόλησε από τότε που μπήκα στην Επιτροπή Ήτρε εδώ και δύο χρόνια. Γιατί δεν βλέπουμε τις πολιτικές κλίματος σε μία νέα πολιτική. Γιατί πολλοί μιλάμε αφενός για τον εμπορικό τομέα, μετά για, τους, για τον μη εμπορικό τομέα. Μπας περιπτώσει θα μπορούσαμε να τους ε, συνδυάσουμε. Μιλάμε και για το πρόγραμμα ε, για τις καύσεις και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποιος, ποιες είναι οι συνολικές επιπτώσεις. Δηλαδή, σε ορισμένους τομείς προχωράμε υπερβολικά πολύ και σε άλλους όχι. Χάνουμε την ουσία δηλαδή πολλές φορές και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον έτσι ώστε να έχουμε συνεκτικές πολιτικές, να μην υπάρχουν επικαλύψεις, να μην, υπάρχουν, να μην υπάρχει υπερβολική ρύθμιση και ούτω καθεξής το ΕΛΚ μίλησε για το 57 και 43%. Εμείς δεν έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα φαίνεται ότι κινηθήκαμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις, δηλαδή ε, θα πρέπει να δούμε ε, κατά πόσο θα πρέπει να πάμε από το μερικό στο γενικό ή αντιστρόφως. Πολλά θέματα βρίσκονται επιτάπητος. Από όλες τις πλευρές θα πρέπει να φτάσουμε σε μία πλειοψηφία. Διαφορετικά δεν θα επηρεάσουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος και το Κοινοβούλιο γενικά. Ας έχουμε λοιπόν μία πολύ διευρυμένη συζήτηση, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε σε μία πλειοψηφία, πλειοψηφική θέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, 6 ώρα το απόγευμα, στις 15 του μηνός Ιουνίου. Μεθαύριο. 6 ώρα το απόγευμα. Tomorrow, voting. Αύριο ψηφίζουμε. Στις 14 του μηνός, 10 η ώρα. Φυσικά συντονιστές ραντεβού στις 9. Γεια σας.